Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. <clears throat> Θα ακολουθήσω την ε, πρόταση του Πολωνού συναδέλφου μου και θέλω να αποτίσω φόρο τιμή σε όλους τους Πολωνούς συναδέλφους που ήρθαν στη συνεδρίασή μας σε μια τόσο πρωινή χρονική στιγμή. Να ευχαριστήσω λοιπόν όλους τους βουλευτές που είναι εδώ παρόντες. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Να σας υπενθυμίσω ότι η συνεδρίασή μας ε, μεταδίδεται στο διαδίκτυο και σε ό,τι αφορά την ερμηνεία οι γλώσσες που έχουν προτεραιότητα είναι οι γλώσσες βέβαια των μονίμων μελών της Προεπιτροπής μας. Θα πρέπει στην αρχή να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Η συνεδρίασή μας θα διαρκέσει δύο μέρες, μία μισή μέρα εν πάση περιπτώσει, μέχρι αύριο το μεσημέρι. Αν δεν έχετε αντιρρήσει ή σχόλια σε σχέση με την ημερήσια διάταξη, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η ημερήσια διάταξη έχει εγκριθεί. τώρα. Έχουμε επίσης την έγκριση των πρακτικών της 3ης Μαρτίου 2016. Εάν μέχρι το τέλος της συνεδριασής μας, λοιπόν, αύριο το μεσημέρι δεν έχουν διατυπωθεί αντιρρήσεις, θα θεωρηθούν τα πρακτικά ότι έχουν εγκριθεί. Περνώ τώρα σε ορισμένε ανακοινώσει της Προέδρου. Αύριο στις 3 ε, στις θα λάβει χώρα μια συνεδρίαση της Επιτροπής ε, Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών της ΙΜΚΟ. Θα λάβει χώρα λοιπόν μια συνεδρίαση που αποτελεί ακρόαση για τα θέματα των δημοσίων αγορών στον τομέα της άμυνας. και θα ήθελα να σας καλέσω να σας ενθαρρύνω να είστε παρόντες στη συνεδρίαση αυτή. Η γραμματεία μας θα σας δώσει και όλες τις αντίστοιχες πληροφορίες και θα τα έχετε όλα αυτά τα στοιχεία σήμερα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Και τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε <clears throat> την συνεδρίασή μας. Έχω την χαρά και την τιμή να παρουσιάσω το πρώτο θέμα της ημερησίας διάταξής μας που είναι η διαμάχη του Ναγκόρνο Καραμπάχ οι επιπτώσεις αυτής της ε, διαμάχης για τη σταθερότητα του Νοτιού Καυκάσου και η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά. Έχουμε λοιπόν μια αντάλλαγη απόψεων με τον ε, ε, ασκούντα τα καθήκοντα του Διευθυντή για την Ρωσία και την Ανατολική Εταιρική Σχέση και την Ευρασία και για τον ΟΑΣΕ την ΟΑΣΕ καλύτερα ο κύριος, είναι ο κύριος Φερνάντο Άντρεσεν Κιμαράις και στη συνέχεια Θα έχουμε την κυρία Αμάντα Πολ του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πολιτικής που είναι ε, <clears throat> αναλυτρία, είναι πεπειραμένη αναλύτρια για τα θέματα πολιτικής ανάλυσης. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα μπορέσει να υπάρξει μια ανακοχή η οποία θα διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα Μετά λοιπόν από την διακεκαυμένη φάση στρατιωτικών επιχειρήσεων μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών, δηλαδή της Αρμενίας και του Αζερβαϊτζάν, σε ό,τι αφορά το ορεινό Καραμπάχ, τον Αγκόνο Καραμπάχ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσοι <coughs> είναι γνωστό, έχει πολλές φορές ασχοληθεί με το θέμα αυτό του Ναγκορο Καραμπάχ. Έχει αναφερθεί σε αυτό και το Κοινοβούλιο σε μια σειρά ψηφισμάτων Έχουμε τονίσει λοιπόν στο παρελθόν και εξακολουθούμε να το πράττουμε και τώρα την ε, αναγκαιότητα του να ληφθούν υπόψη σε μια κατάσταση όπως αυτή τα θέματα της εδαφικής ακαιρεότητος των κρατών της περιοχής και θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκυμαράης και την κυρία Πολ και μετά θα μπορείτε να θέσετε ερωτήματα ή να κάνετε σχόλια. Επειδή η κυρία Πολ θα πρέπει να αποχωρήσει νωρίτερα, ε, δίνω το λόγο καταρχήν στον κύριο Κιμαράης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα. Πράγματι, η πρόσφατη κλιμάκωση της βίας ε, στις αρχές Απριλίου, όπως αναφέρεται, αποδεικνύει ότι αυτή η διαμάχη του Ναγκόνο Καραμπάχ δεν είναι παγωμένη και πράγματι η κατάσταση παραμένει ασταθής στην περιοχή. Αστάθεια η οποία αποτελεί απειλή για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής και των γύρω περιοχών. Όπως ανέφερε η κυρία Μογκερίνη, αυτή η διαμάχη παρεμποδίζει την ανάπτυξη και τη σταθερότητα των δύο χωρών, των γειτονικών χωρών και τις σχέσεις τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κάνει έκκληση πολλές φορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να εντείνει το ρόλο της ώστε να τερματιστεί η διαμάχη στην περιοχή και πρόσφατα η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος υποσχέθηκε να εργαστεί για αυτό το σκοπό. Οι στόχοι της ανατολικής γειτονίας μπορούν να επιτευχθούν μόνο με τη σταθερότητα στην περιοχή. Η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος λοιπόν επισκέφθηκε το Αζερμπαϊτζάν τέλη Φεβρουαρίου και την Αρμενία αρχές Μαρτίου για συναντήσεις αντίστοιχα με τους Προέδρους και Υπουργούς Εξωτερικών των δύο χωρών αυτών τους παρότρινε για ε, να προχωρήσει η ειρηνευτική διαδικασία. Αυτά τα μηνύματα που επαναλαμβάνει και ο κύριος Σάμπα στις τακτικές του συναντήσεις ε, ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με τους υπουργούς αυτών των χωρών. Όσον αφορά την κρίση αρχές Απριλίου, μετά από μια νύχτα συγκρούσεων, η εκπρόσωπος έκανε έκκληση για διακοπή των εχθροπραξιών και αποχή από τη χρήση βίας. Το κατά πόσο θα γίνουν περισσότερα θα εξερθεί από τη βούληση των δύο πλευρών να αποδεχθούν περισσότερο το δικό μας, ε, τη δική μας συμμετοχή και τις δικές μας συμβουλές. Άμεση προτεραιότητα αποτελεί η διασφάλιση της ε, τήρησης τη συμφωνία ε, Παύσης πυρό. και πρέπει να επιμένουμε ότι η λύση για αυτή τη διένεξη είναι μόνο πολιτική. Η στρατιωτική επιλογή πρέπει να απορριφθεί και από τις δύο πλευρές. Συνεπώς είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλήσει με μία φωνή όσον αφορά την υποστήριξη της ομάδας Μίνσκ του ΩΣΑ ε, που είναι ο διεθνής οργανισμός που έχει συμφωνηθεί για τη διαθέτηση αυτής της διαμάχης. Και στο πλαίσιο αυτό της εργασίας των συμπροέδρων ε, της ομάδας Μίνσκ υπάρχει ανάγκη να επανεκκινηθούν οι διαπραγματεύσεις σε βάση των αρχών της Μαδρίτης. Τη μη χρήση βίας ε, την τήρηση της εδαφικής ακυριότητας και το δικαίωμα αυτοδιάθεσης. Σε αυτές τις διαπραγματεύσεις ε, και οι δύο πλευρές πρέπει να είναι έτοιμες ε, για ε, διαπραγματεύσεις αποτελεσματικές βασισμένες σε αμοιβές υποχωρήσεις. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό να παραμείνει η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ενταθούν οι πολιτικές προσπάθειες για τη διευθέτηση της διένεξης και να δοθούν μηνύματα για την οικοδόμηση της ασφάλειας συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός μηχανισμού έρευνας περιστατικών όπως προτείνεται από τον ε, ΟΑΣΕ και τον οποίο έχει υποστηρίξει ρητά και η κυρία Μογκυρινίδη. Μαζί με την τήρηση της εκεχηρίας και τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που θα βοηθά την πρόοδο. Οποιασδήποτε δηλώσεις και δράσεις που περιπλέκουν περαιτέρω το ήδη περίπλοκο περιβάλλον πρέπει να σταματήσουν. Είναι σημαντικό να στείλουμε ισόρροπα μηνύματα και όχι μεροληπτικά υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την επίσημη ειρηνευτική διαδικασία μέσω των δραστηριοτήτων της υπέρ εκπροσώπου και του εκπροσώπου ε, κ. Σάμπα με επαφές ε, ε, και στις δύο πλευρές της διαμάχης. Ο κ. Σάμπα ταξίδευσε στο Αζερμπαϊτζάν την περασμένη εβδομάδα στι 15 Απριλίου και σύντομα πρόκειται να επισκεφθεί την Αρμενία. Στο Αζερμπαϊτζάν συνάντησε τον Πρόεδρο, τον Υπουργό Άμυνα και τον Υπουργό Εξωτερικών και την ίδια μέρα συνομίλησε δύο φορέ με τον Αρμένιο Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίο βρισκόταν σε επίσκεψη στην Κίνα διότι η επίσκεψη ε, στην Αρμενία δεν ε, ήταν δυνατόν να λάβει χώρα λόγω της ε, απροσδόκητης απεργίας στο αεροδρόμιο Ζάβαντα των Βρυξελών. Αλλά θα γίνει σύντομα. Ο κύριος Σάμπα εξακολουθεί να είναι σε στενή επαφή με τους συμπροεδρούς της ομάδας Μίνσκ με τακτικές τηλεφωνικές συνομιλίες. Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τις ε, δραστηριότητε οικοδόμηση τη Ειρηνή και έχει και επαφέ με διάφορου ανθρώπου όπως ανέφερα και με το πρόγραμμα Ευρωπαϊκή Εταιρική Σχέση για τη Διευθέτηση ειρηνικά της διαμάχης των Αγκονοκραμπάχ. Τα προγράμματα αυτά ε, βοηθούν στις επαφέ μεταξύ ανθρώπων και αποτελούν μια απόπειρα γεφύρωσης των διαφορών. Εμείς θεωρούμε ότι τα μέτρα οικοδόμησης της εμπιστοσύνης θα, θα παίξουν ουσιώδη ρόλο για την ε, μακροχρόνια συμφιλίωση και μπορούν να υποστηρίξουν την πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Βάσει των αρχών της Μαδρίτης, ε, η λύση θα βρίσκεται τελικά στα χέρια των δύο μερών της διάνεξης, αλλά πρέπει και οι δύο να κάνουν συμβασμούς ε, υπέρ της ειρήνης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Διευθύντα. Θυμίζω ότι ε, εκτελεί χρέη ε, διευθυντού ο κύριος Γκυμαράης στην ΠΙΕΔ. Και τώρα η κυρία Αμάντα Πολ, πολιτική αναλύτρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πολιτικής. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση σήμερα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να υπερεκτιμήσουμε τη σοβαρότητα της ε, πρόσφατης κλιμάκωσης της βίας στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Ήταν η σοβαρότερη κλιμάκωση από το 1994. Περισσότεροι άνθρωποι σκοτώθηκαν αυτές τις μέρες από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Συμπεριλαμβανομένων μικρών παιδιών, πολλοί επίσης εγκατέλειψαν τα χωριά τους ε, παράλληλα με τη γραμμή επαφής και αυτό είναι πολύ λυπηρό. Καταρχήν η κλιμάκωση αυτή ήταν τελείως προβλέψιμη γιατί αν δείτε τα προηγούμενα κάνα δύο χρόνια υπήρχε αύξηση των συγκρούσεων σοβαρών το Νοέμβριο του 2014, το Δεκέμβριο του 2015 υπήρξε και τερά... υπήρχαν πάρα πολλές στρατιωτικές ασκήσεις στο Αζερβαϊτζάν και στα κατεχόμενα εδάφη κοντά στη γραμμή επαφής. Είναι προβλέψιμο επίσης ότι θα συμβεί ξανά κλιμάκωση της βίας. Το βασικό ερώτημα είναι πότε θα γίνει η κλιμάκωση. Μια άλλη προβλεψιμότητα ήταν ο πολύ ενεργός ρόλος της Ρωσίας. Δεν εκπλήσει ότι οι Ρώσοι πήγαν να βοηθήσουν διότι άρχισαν σε μαζική κλίμακα μια πρωτοβουλία. Τα επεισόδια έγιναν όταν οι δύο πρόεδροι έλειπαν στην Ουάσιγκτον και αυτό πραγματικά ήταν πολύ σημαντικό και σοκάρι αρχίζουμε νέα φάση στη σύγκρουση, γιατί το καθεστώς που προϋπήρχε ε, συνετρίβει, δεν μπορούμε να ξαναγυρίσουμε σε αυτό, αποτελεί παρελθόν. Και νομίζω ότι όταν μιλάμε για κατάπαυση του πυρός υπό τις παρούσες συνθήκες, αυτό είναι λίγο αστείο, γιατί παρά το γεγονός ότι οι Ρώσοι διαπραγματεύτηκαν νέα κατάπαυση του πυρός, βλέπουμε ότι από τότε, δηλαδή λίγες μέρες πέρασαν μόνο από τότε, υπήρξαν εκατοντάδες παραβιάσεις. Οπότε ήδη βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη ενδιαφέροντος για τη νέα κατάπαυση του πυρός και κανείς δεν θέλει να εφαρμοστεί πλήρως. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πολύ ασταθή και αβέβαιη ε, κατάσταση και επικίνδυνη δυναμική επιτόπου. Μπορεί δηλαδή να συνεχίσουν να αναπτύσσονται δυνάμεις και των δύο πλευρών. Τώρα, για την ίδια τη σύγκρουση δύο λόγια. Καταρχήν το Καραμπάχ δεν μοιάζει με τις άλλες συγκρούσεις της περιοχής που τις ονομάζουμε παγωμένες. Όπως ακούσαμε, δεν είναι παγωμένη σύγκρουση και ποτέ δεν ήταν. Από το 1994 υπήρχαν συνεχείς παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός. Αλλά με, το, με τα χρόνια γίνονταν πιο σοβαρές. Ε, πέρασαν οι καιροί των ε, περιστασιακών ε, συγκρούσεων. Τώρα η σύγχρονη τεχνολογία, ο στρατιωτικός εξοπλισμός που απέκτησαν και οι δύο πλευρές άλλαξαν τα δεδομένα. Αυτή η περιοχή τώρα είναι πλέον στρατιωτικοποιημένη στην ευρύτερη Ευρώπη. Δισεκατομμύρια έχουν δαπανηθεί για σύγχρονα όπλα, ε, τάγκ, βαρύ πυροβολικό, ε, μη επανδρομένα ε, ροσκάφη. 4,6% του ΑΕΠ του Αζερβαϊτζάν πάει στον αμυντικό προϋπολογισμό και 4,1% του αρμενικού προϋπολογισμού. Το ΑΕΠ των δύο χωρών διαφέρει πολύ, αλλά παρόλα αυτά μιλάμε για μεγάλα κονδύλια ε, που δαπανώνται στα, στους εξοπλισμούς. Η Αρμενία παίρνει τα περισσότερα όπλα από τη Ρωσία και το Αζερβαϊτζάν από το Ισραήλ, Τουρκία, Ρωσία και από το Πακιστάν επίσης όπως πιστεύουν πολλοί. Ε, επίσης ε, υπάρχει η στρατηγική ε, εταιρική σχέση Αρμενίας-Ρωσίας και συμφώνησαν πρόσφατα ε, πωλήσει ε, σε αρχές του χρόνου ύψους 200 εκατομμυρίων. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι τώρα οι εθνικιστές και στις δύο πλευρές έχουν ισχυρότερο λόγο. Οι Αρμένοι και οι Αζέροι θεωρούν ο ένας τον βασικότερο εχθρό του άλλου. Και αυτό είναι σημαντικό. Πριν από 35 χρόνια δε συμβίωναν ε, φιλικά οι δύο λαοί. Ε, οπότε αυτή η αλλαγή έγινε από τις δύο ηγεσίε. Τώρα η κατάσταση διαμορφώθηκε από διάφορα στοιχεία. Καταρχήν υπήρχε κολλησιεργία στην ειρηνευτική διαδικασία και δεν έγιναν σημαντικές συναντήσεις μεταξύ των δύο ηγετών για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Πράγμα που σημαίνει ότι η ομάδα του Μίνσκ έγινε ουσιαστικά ένας μάνατζερ μάλλον παρά επιλητή προβλημάτων. Επίσης η εμπιστοσύνη μεταξύ Ρωσίας και Δύσης ε, μειώθηκε και αυτό επιδεινώθηκε και από την Ουκρανική σύγκρουση που θεωρήθηκε και από την Αρμενία και από το Αζερμπαϊτζάν με διαφορετικούς τρόπους και το συνεχιζόμενο ε, πρόβλημα της παρακολούθησης επιτόπου. Ε, υπάρχει μια ομάδα οκτώ ε, ανθρώπων που παρακολουθούν τις εξελίξεις, περιορισμένη ομάδα και μπορούμε να πούμε ότι είναι αναποτελεσματική. Η σημερινή κατάσταση, ε, το, το σημερινό καθεστώς είναι πιο ευνοϊκό για την Αρμενία από ότι για το Αζερβαϊτζάν, γιατί είναι προφανές ότι υπάρχει η πεποίθηση ότι στο βαθμό που υπάρχει αυτή η κατάσταση είναι πιο πιθανό να αναγνωριστεί τον Αγκόρνο Καραμπάχ ως ανεξάρτητο κράτος. Γενικά και οι δύο χώρες θα έλεγα ότι ασχολήθηκαν περισσότερο ε, μία κατά της άλλης παρά αναζητώντας συμβιβαστική λύση ε, και ε, την πιθανότητα να αποκομίσουν αμοιβαία ωφέλη. Και αυτό αξιοποιήθηκε και από τις δύο πλευρές ε, για να αποσπάσουν την προσοχή του πληθυσμού από άλλα σοβαρά εσωτερικά θέματα. Ε, τώρα, αν δούμε τα επεισόδια που άρχισαν στις 2 Απριλίου, τι έγινε εκεί. Πρόκειται για δύο δυνα... πιθανότητες. Πρώτα απ' όλα, ε, σταμάτησε να ισχύει η κατάπαυση του πυρός και μετά κλιμακώθηκε η κατάσταση ε, μετά από ε, δυσμενείς εξελίξεις στο προηγούμενο διάστημα. Οι Αζέροι ακούμε ότι αποφάσισαν να κάνουν μια ε, ταχεία σύντομη στρατιωτική επιχείρηση για να αλλάξουν τα δεδομένα επιτόπου και να δοκιμάσουν καινούριο όπλα και να εφαρμόσουν μια νέα στρατηγική που ορισμένοι ε, θεωρούν και χαρακτηρίζουν ως ε, ασφαλή στρατηγική για να ανακτήσουν κάποιες κατεχόμενες περιοχές. Ως ένα βαθμό νομίζω ότι το Αζερμπαϊτζάν έχει απογοητευθεί διότι επί δύο δεκαετίες ε, εδάφη του είναι κατεχόμενα, τα ψηφίσματα του ΙΕ αγνοούνται και η ειρηνευτική διαδικασία δεν οδηγεί πουθενά. Και υπάρχει ε, περιορισμένη, ε, περιορισμένο ενδιαφέρον από τη Δύση και την Ευρωπαϊκή Ένωση. βέβαια θεωρούν ότι η χρήση των όπλων δεν είναι παραδεκτή. Αν δούμε όμως τώρα την κατάσταση, στο Αζερμπαϊτζάν υπάρχει μια αίσθηση νίκης, γιατί για πρώτη φορά ε, ανέκτησε εδάφη από τότε που συμφωνήθηκε η κατάπαυση του πυρός το 1994. Παράλληλα όμως το γεγονός ότι το Αζερμπαϊτζάν δεν επίεσε για να αποκτήσει ολόκληρη την περιοχή, αυτό δείχνει ότι η αρμενική αντίδραση ήταν αρκετά αποτελεσματική. αλλά η κατάσταση παραμένει αβέβαιη. Υπάρχουν τρεις ε, εναλλακτικέ τώρα ε, επιτάπητος. Πρώτον, η καλύτερη λύση θα ήταν να επιστρέψουν στις διαπραγματεύσεις για μια συνολική επίλυση στα πλαίσια των αρχών της Μαδρίτης. Η δεύτερη εναλλακτική είναι να γίνει νέα κλιμάκωση τις επόμενες εβδομάδες και μήνες και θα είναι πιο καταστροφικές οι συνέπειες από ό,τι αυτές που είδαμε. Και η τρίτη, και αυτό με ξαναγυρίζει στους Ρώσους, το σχέδιο που προχωρούν οι Ρώσοι και το συζητούν με διάφορα μέρη, θα εφαρμοστεί κατά κάποιο τρόπο από τα μέρη και έτσι θα γίνει εγγυήτρια της ειρήνης επιτόπου η Ρωσία. Αυτό είναι το λιγότερο πιθανό, αλλά ε, παραμένει εναλλακτική. Και πιστεύω ότι ε, αν δεν υπάρξει άμεση επιστροφή στην πολιτική διαδικασία, είναι πιθανό να πιεστεί το Αζερβαϊτζάν να προχωρήσει σε νέα επίθεση ή να δεχτεί την ε, συμφωνία των Ρώσων. Γιατί στο τέλος μπορεί να πούν ότι καλύτερα να συμφωνήσουμε με τους Ρώσους για να ξαναπάρουμε κάποια κατεχόμενα παρά να συνεχίσουμε ε, σε μια διαδικασία που δεν οδηγεί πουθενά. Τώρα, δύο λόγια επίσης για τη Ρωσία. Ε, και τη ε, διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να δούμε προσεκτικά τι κάνουν οι Ρώσοι στην περιοχή, γιατί δεν είναι ειρηνοποιός η Ρωσία. Ε, για χρόνια ε, πολλούσε όπλα και έτσι αναζωπήρωνε την σύγκρουση. Το, αυτό δεν βοηθάει το Αζερμπαϊτζάν και τη Ρωσία. Ο πρόεδρος Βέγεφ είπε ότι δεν θα σταματήσουν να πολλούν όπλα, γιατί πιστεύουν ότι και μέλη του ΝΑΤΟ εξακολουθούν να ε, θα, θα, παρέμβουν και θα πουλήσουν. Ο βασικός στόχος της Ρωσίας είναι να ελαχιστοποιηθεί η πολιτική επιρροή άλλων σε αυτή την περιοχή, γιατί πιστεύουν ότι είναι επιτακτικό να είναι η κυρίαρχη δύναμη ε, στο Νότιο Κάφκασο και στη σύγκρουση αυτή. Και αν δούμε τα βήματα της Ρωσίας μετά την κλιμάκωση, ήταν η πρώτη η Ρωσία που αντέδρασε στα επεισόδια της Δευτέρας Απριλίου. Μετά ο πρόεδρος Πούτιν έκανε ε, μια δήλωση και ε, επικοινώνησε ε, με τους υπουργούς άμυνας και εξωτερικών με του Αζερβαϊτζάν και της Αζερβαϊτζάν Αρμενίας και ο Λαυρόφ πήγε στις δύο χώρες. Και ε, αν σκεφτούμε μελλοντική ρωσική συμφωνία, θα, αυτή θα σημαίνει επιστροφή των κατεχομένων, ε, θα είναι η ειρηνευτική δύναμη Ρώση και θα υπάρχουν κάποιες εγγύσεις ε, ασφάλειας για τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Ε, οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν λίγα στοιχεία των αρχών της Μαδρίτης. Η, Ρώσοι ε, που θέλουν οι Ρώσοι να περάσουν ε, στα πλαίσια του ΟΑΣΕ. Νομίζω ότι εξακολουθεί να είναι δύσκολη η κρίση και ε, ίσως η λύση αυτή δεν θα είναι δημοφιλή στην περιοχή. Η Τουρκία επίσης είναι ε, εναντίον γιατί δεν θέλει να περικυκλωθεί από ρωσικές ειρηνευτικές δυνάμεις η Τουρκία. Δεν μπορώ να φανταστώ δηλαδή ότι θα ικανοποιηθούν. Επίσης ε, ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι η Δύση δεν φαίνεται να ανησυχεί πολύ για τη θέση που παίρνει στην περιοχή η Ρωσία που ενισχύει τη θέση της και σε σχέση με τη σύγκρουση και σε όλο τον Κάφκασο. Αυτό είναι λάθος. Η Δύση, ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού είναι ο πιο κοντινός παίκτη, ε, σε μια εποχή όπου οι Αμερικανοί ε, απομακρύνονται λόγω της ε, προεκλογικής διαδικασίας δεν θα παίξει σημαντικό ρόλο δηλαδή ο πρόεδρος Ομπάμα αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να το κάνει διότι αυτά που συμβαίνουν εκεί έχουν άμεσο αντίκτυπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταρχήν πρόκειται για νέα, ε, ε, μια νέα σύγκρουση, μπορεί να ξεπεράσει τα σύνορα αυτή τη περιοχή, μπορεί να δημιουργήσει νέο κύμα προσφύγων, μπορεί να βλάψει ε, κέρυε υποδομέ. Μέχρι τώρα υπήρξε έλλειψη πολιτικής βούλησης πολλών από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξουν σημαντικό ρόλο στα πλαίσια του ΟΑΣΕ. Και αν δείτε την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε άλλες, ε, στη Γεωργία, στην Υπερδινιστερία, ε, είναι πολύ πιο ε, προορατική προσέγγιση. Αυτό δεν συμβαίνει στον Αγκόρνο Καραμπάχο, που υπάρχει έλλειψη στρατηγικής επένδυσης. Και νομίζω ότι υπάρχει μία χαλάρωση, θεωρώντας ότι θα σταματήσει η σύγκρουση. Όμως ε, είναι σημαντικό ε, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της κυρίας Μογκερίνη ε, στις αρχές του χρόνου ε, υπογραμμίστηκε ότι το Ναγκόρνο Καραμπάχ πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι πολύ θετικό. Είναι σωστή προσέγγιση, πιστεύω. Ε, τώρα, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πολιτικής, ε, ε, ένα συνάδελφος και εγώ έχουμε καταρτήσει ένα κείμενο για τον Αγκόρνο Καραμπάχο, που έχουμε καταγράψει κάποιες ιδέες για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βελτιώσει την προσέγγιση της και να παίξει σημαντικότερο ρόλο. Καταρχήν πρέπει να πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και χαιρετίζω το γεγονός ότι εσείς αναλάβατε πρωτοβουλία σε πολλές περιπτώσεις και παρουσιάσατε ιδέε για να ενισχύσετε τον ρόλο τη Ένωση στην περιοχή. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Είναι το μοναδικό θεσμικό όργανο τη της που το έχει κάνει αυτό. Να πω κάποια πράγματα που καταγράψαμε εγώ και ο Ντένις. Καταρχήν είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εκπροσωπείται ε, ε, περισσότερο στα πλαίσια της ομάδας του Μίνσκ, είναι πολύ σημαντικό αυτό, ε, στην ευρύτερη ομάδα, όχι, όχι ο συμπρόεδρος. Και Παράλληλα, είναι σημαντικό να συμμετέχει η ομάδα του Μίνσκ χρειάζεται περισσότερη σκέψη, περισσότερες χώρες που θα συμμετέχουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επίσης να θεωρήσει το Καραμπάχ ως σημαντικό κομμάτι του πολιτικού διαλόγου και με την Αρμενία και με το Αζερβαϊτζάν και να μην το παρακάμψει, πράγμα που συνέβη μέχρι τώρα. Επίσης προτείνουμε ότι ε, θα πρέπει να ορίσει στρατιωτικούς ε, αξιωματικούς συνδέσμους ε, και στο Πακού και στο Γεριβάν. Θα πρέπει να συνεχίσει να συμμετέχει μέσα από την κοινωνία των πολιτών με το EPNK ε, είναι κρίμα που χρειάστηκε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα για να αρχίσει η χρηματοδότηση του PNK. Ε ε, δεν ξέρω γιατί συνέβη αυτό, αυτή η καθυστέρηση, αλλά είναι κρίμα διότι η διπλωματία και η διαμεσολάβηση είναι κέρια σημασίας. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διασφαλίσει περισσότερο ότι θα είναι πιο συγχρονισμένες οι κινήσεις για το Καραμπάχ, γιατί τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικές θέσεις, θα πρέπει να συγχρονίσουν λοιπόν, να, να συντονίσουν την άποψή τους, και αυτό, γιατί η διασπορά απόψεων και η διαφορά δεν βοηθάει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει και η Πρόεδρος και τους δύο μιλητές μας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Ο κύριος Κέλαμα έχει το λόγο καταρχήν από την ομάδα του ΕΡΚ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους ομιλητές μας για την ενημέρωση και τις πληροφορίες που μας έδωσαν για αυτό το αρκετά πολύπλοκο πρόβλημα. Όπως ε, μόλις είπατε, έχει ανατραπεί το status quo στην περιοχή, αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Δεν πρέπει να τρέφουμε ελπίδες ότι μπορούμε απλώς να επανέλθουμε στην προηγούμενη επισφαλή κατάσταση. Το βασικό ερώτημα εδώ το οποίο τίθεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ποιος εποφελείται από τέτοιες διαμάχες. Πριν από τρία χρόνια, πριν από, συγγνώμη, 90 χρόνια, το 1923, ο Στάλιν αποφάσισε να δώσει τον αγκόνο Καραμπάχ στο Αζερβαϊτζάν ενώ ήταν μια περιοχή κυρίως με αρμενικό πληθυσμό. Αυτή ήταν ε, η σπορά των ε, συγκρούσεων, αν θέλετε, που έγινε τότε, χρησιμοποιώντας τη λογική του «διέρη και βασίλευε». Αλλά αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό και για την Αρμενία και για το Αζερβαϊτζάν. Η σχέση της Αρμενίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παγώσει λόγω αυτής της κατάστασης οι εντάσεις αυτές την έχουν κάνει να παραμελήσει σημαντικά προβλήματα οικονομικής ανάπτυξης στην Αρμενία. Το Αζερμπαϊτζάν πηγαίνει όλο και χειρότερα σε ό,τι αφορά τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η σύγκρουση αυτή στον Αγκόρο Καραμπάχ είναι ένα πολύ καλό πρόσχημα για να αφαιθούν τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην άκρη. Το ερώτημά μου είναι σε σχέση με τον δυνητικό ρόλο της γεωργίας στην ε, σύγκρουση αυτή. Θα μπορούσε η Γεωργία να διαδραματίσει κάποιο ρόλο. Είπατε επίση ότι οι σχέσεις του Αζερμπαϊτζάν με το Ιράν είναι σημαντικέ. Ενδιαφέρεται το Ιράν πράγματι ενεργά για αυτή τη διαμάχη ή όχι. Και το τελικό συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει μια έλλειψη ενεργού και δυναμικού ρόλου της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Έχουμε αφήσει τα θέματα αυτά να τα κάνει η Ρωσία όπως θέλει και φαίνεται ότι θα γίνει δεκτή η πρόταση της τη Ρωσία τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποια άλλη εναλλακτική λύση. Σας ευχαριστώ. Ο κύριο Πάσκου έχει το λόγο. Και εγώ θέλω να σα ευχαριστήσω για την ε, συζήτηση αυτή που είναι ιδιαίτερα επίκαιρη γιατί όλοι μας έχουμε ανησυχήσει με την ένταση και την ταχύτητα με την οποία ξέσπασε η βία και πάλι στην περιοχή του Ναγκόνο Καραμπάχ. Ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει αυτή η υποβόσκουσα σύγκρουση, το έχουμε αντιμετωπίσει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά δεν έχουμε δώσει πάντα την απαιτούμενη προσοχή. Και ούτε και τα πιο εκτελεστικά κομμάτια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αντιμετωπίσει το θέμα αυτό. Σαν τα ηφαίστεια, ποτέ δεν ξέρει κανείς πότε είναι η επόμενη έκρηξη ενός ηφαιστείου. Γι' αυτό πιστεύω θα πρέπει να παρακολουθήσουμε από κοντά και συνεχώς να παρακολουθούμε αυτήν την κατάσταση. Πολλές φορές υπάρχουν συγκρούσεις οι οποίες εμφανίζονται σε περιοχές που είναι ειρηνικές και δεν τις περιμένει κανείς. Αλλά εδώ μια τέτοια ανασωπήρωση της βίας είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να το περιμένουμε. Είναι απαραίτητο λοιπόν να έχουμε μια συνεχή εποπτεία αυτών των καταστάσεων. Όπως και άλλες διαμάχες, αυτή η διαμάχη έχει το ορατό κομμάτι, τους ορατούς εμπλεκόμενους και μετά υπάρχουν αυτοί οι οποίοι είναι η μη ορατή, η Τουρκία, η Ρωσία, ίσως το Ιράν. Δεν ξέρω αν αυτό είναι τμήμα μιας γενικής ε, υποβάθμισης των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας. Ίσως κάπως μπορεί να συναρμοστεί σε ένα τέτοιο υπόδειγμα, αλλά υπάρχει και ένα άλλο ορατό στοιχείο αυτής της κατάστασης. Σήμερα τίθεται το θέμα της ελευθερίας έκφρασης από την πλευρά των ε, δεξαμενών σκέψης και η αυτοσυγκράτηση που πρέπει να κρατήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια ένταση μεταξύ των δύο αυτών θέσεων. Αλλά εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε να ασχοληθούμε μόνο με τους άμεσα εμπλεκόμενους γνωρίζοντας ότι δεν είναι αυτοί οι οποίοι θα έχουν τον τελικό λόγο για το πώς θα εξελιχθεί αυτή η διαμάχη έχουμε την ευκαιρία να δείξουμε ότι κάνουμε κάτι, ότι μιλάμε για την ανάγκη να υπάρχει επαφή μεταξύ των δύο πλευρών που θα είναι η καλύτερη λύση σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Ξέρουμε ότι αυτό δεν γίνεται γιατί οι πραγματικά εμπλεκόμενοι αυτοί που κουνούν τα νήματα πίσω από την σκηνή Ρωσία, το Ιράν, η Τουρκία και όλοι αυτοί είναι πάρα πολύ ενεργοί και αυτοί αποφασίζουν για τα τεκτενόμενα. Μήπως λοιπόν θα πρέπει να θίξουμε αυτό το θέμα όταν συζητήσουμε, όταν συναντηθούμε με τη Ρωσία ή με την Τουρκία και να συζητήσουμε για αυτά τα ζητήματα πιο σοβαρά. Ξέρω ότι μπορούμε πάντα να είμαστε ικανοποιημένοι με τον χαμηλότερο κοινό παρονομαστή, ότι έχουμε κάνει κάτι στην ομάδα του Μίνσκ, ότι έχουμε αναφερθεί στις αρχές της Μαδρίτης, έχουμε τονίσει την ανάγκη να υπάρχουν επαφές μεταξύ των δύο πλευρών σε επίπεδο απλών ανθρώπων, αλλά μπορεί να περιοριστούμε μοναχά σε αυτά και την επόμενη φορά θα ξαναγίνουν τα ίδια. Και νομίζω ότι η κυρία Πολ τόνισε και εξήγησε πολύ καλά ότι υπάρχει δυνατότητα αυτή η διαμάχη να οξύνει ακόμα περισσότερα τα προβλήματα τα οποία έχουμε στην περιοχή του Νότιου Καυκάσου. Μπορεί αυτό να συνδεθεί με την κατάσταση στο Ιράκ και τη Συρία ή με άλλε περιοχέ. Γι' αυτό πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή και να απευθυνθούμε στου πραγματικού ε, εμπλεκόμενους σε αυτή την ε, περίπτωση και δεν ξέρω αν μπορείτε να μου βοηθήσετε προ την κατεύθυνση αυτή. Ο κύριος Μάρεκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους για τις πολύ σημαντικές και ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Να ευχαριστήσω ειδικότερα την Πρόεδρο που οργάνωσε αυτή τη συζήτηση σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Η υποεπιτροπή μας ε, έχει σημαντικό ρόλο, οπότε πρέπει να ε, αντιδράσει ε, γρήγορα. Θα ήθελα να σας κάνω μερικές ερωτήσεις όσον αφορά την Τουρκία και την Αρμενία. Η θέση του Αζερβαϊτζάν, η ε, πολιτική της Τουρκίας, υπάρχει μια εθνική αλληλεγγύη. Υπάρχουν κάποιες ευρύτερες προοπτικές γεωπολιτικές στην τουρκική πολιτική αυτό που θα ήθελα λοιπόν να μάθω είναι αν ε, έχει αλλάξει πολιτική ο Ερντογάν όσον αφορά την Αρμενία. Θα ήθελα να μάθω ποια είναι η θέση της Αρμενίας όσον αφορά τη Ρωσία. Όπως ξέρουμε η Ρωσία υπερασπίζει την θέση της Αρμενίας ε, ε, η οποία βρίσκεται σε σημαντική γεωπολιτική θέση. Θέλαμε λοιπόν να μαθούμε αν η θέση των αρμενικών αρχών είναι εξαρτώμενη από τις θέσεις της Ρωσίας ή αν απλά έχουν κάποια σχέση ε, θετική, καλή, ας, πούμε, ας το πούμε έτσι. Επίσης, ε, όσον αφορά την θέση εντός της Αρμενίας, ε, εμείς ε, ως ε, δυτική δύναμη μπορούμε να κάνουμε κάτι, να αυξήσουμε την παρουσία μας ε, ώστε να βοηθήσουμε στη σταθερότητα της περιοχής. Μήπως καταφέρουμε να δώσουμε και μια λύση στο διένεξη ο κύριος Μαυρίδης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τρεις σύντομες παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω και θα ήθελα να έχω την ε, απάντηση των καλεσμένων μας. Θα ήθελα καταρχήν να επαναλάβω αυτά που είπε η ύπατη εκπρόσωπος Μογκερίνη στο Στρασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα. Το έκανε απόλυτα σαφές ότι με στρατιωτικές αντιπαραθέσεις όπως αυτή του Ναγκόρνο Καραμπάχ δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε πολιτική λύση του του βέβαια. Καταρχήν θα πρέπει να σκεφτούμε τη δική μας θέση ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρω ότι η ηθική δεν συμβαδίζει με την πολιτική. Είμαι από την Κύπρο και το έχω δει αυτό στις σχέσεις μας με την Τουρκία. Πολλές φορές όμως πιστεύω ότι υπάρχει μια πραγματική διαφορά μεταξύ του να είναι κανείς πεπισμένος, πεπισμένος για το δίκιο του και του να είναι απλώς ουδέτερος. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να κρατήσουμε μια αμερόληπτη και ουδέτερη στάση και να πούμε τα πράγματα όπως είναι. Και έρχομαι στο επόμενο σημείο που θέλω να δείξω. Χρειαζόμαστε ίσως, μήπως χρειαζόμαστε ένα αποτελεσματικό μηχανισμό που θα βοηθήσει και τους Αρμένιους και τους Αζέρους και θα σώσει ανθρώπινες ζωές. Ναι, είναι η απάντηση δική μου. Χρειάζεται κάτι τέτοιο. Μία πρόταση, κάτι κάποια προσπάθεια μέσω της ομάδας του Μίνσκ όπου υπάρχει και η Ρωσία και η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες και έχουν πραγματικά προτείνει κάτι. Εγώ πρέπει να πω ότι σε αυτή την περίπτωση βλέπω να το έχει δεχτεί αυτό τη μεσολάβηση της ομάδας του Μίνσκ και η Αρμενία αλλά όχι το Αζερμπαϊτζάν. Τώρα, όπως έχει λεχθεί από ένα από τους συναδέλφους μου, ένα από τα βασικά ερωτήματα, όπως είπε ο κ. ποιος είναι αυτός ο οποίος επωφελείται από αυτή την κατάσταση πέραν των εμπορών όπλων, των χωρών που πουλούν όπλα όπως η Ρωσία. Ας δούμε τις δύο αυτές χώρες. Να το αναδιατυπώσω. Ποιος είχε κίνητρο αυτή τη φορά να υπάρξει και πάλι μια επιθετική ενέργεια, η οποία οδήγησε στην ε, αναζωπήρωση της σύγκρουσης. Και νομίζω το ξέρουμε όλοι. Θα ήθελα να έχω την απάντηση των καλεσμένων μας για το θέμα αυτό. Είναι κάτι το οποίο οφείλεται σε εσωτερικά προβλήματα λόγω της οικονομικής δυσπραγίας στο Αζερβαϊτζάν. Υπάρχει μια προσπάθεια το Αζερβαϊτζάν να κοροϊδέψει το λαό του μέσω αυτής της ε, διαμάχης ή όχι. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Νικολάη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να σας συγχαρώ πρώτα απ' όλα που επιλέξατε αυτό το σημείο προς για σήμερα. Για μένα είναι πολύ σημαντικό. Εγώ είμαι η συγγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Αζερμπαϊτζάν και ήθελα επίσης ε, να συγχαρώ και τους ομιλητές ε, για την πολύ ισορροπημένη προσέγγιση του ζητήματος. Για μένα το πρόβλημα είναι ποιος θέλει ειρήνη και ποιος θέλει πόλεμο. Πιστεύω ότι έχουμε έναν εκεί στην περιοχή που θέλει να κάνει πόλεμο και κάποιες φορές ε, παίζει το ρόλο του ειρηνευτή ε, και αναφερόμαστε στο προφανή υποπτώ τη Ρωσία διότι η Ρωσία ενδιαφέρεται να διατηρεί αυτές τις προνομαζόμενες παγωμένες συγκρούσεις όπως και να τις ονομάσουμε οι διαμάχες είναι υπαρκτές έχουμε πολλές παγωμένες συγκρούσεις ε, στην περιοχή έχουμε την Απχαζία όχι μόνο τον Κάφκασο και οι παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός ξεκινούν στη συγκεκριμένη περίπτωση διότι η οικονομία του Αζερμπαϊτζάν δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση λόγω της τιμής του πετρελαίου. Το πρώτο θύμα αυτών των παραβιάσεων είναι πολίτες του Αζερμπαϊτζάν που ζουν κοντά. Αυτοί υποφέρουν από τις βιοπραγίες. Ε, γιατί από την άλλη πλευρά του Ναγκοροκαραμπάχ δεν υπάρχουν, δεν κατοικούν πολίτες. Για μένα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό, διότι πρέπει να έχουμε μια ρεαλιστική άποψη ε, για θέματα διεθνούς δικαίου. Έχουμε τέσσερα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Δεν έχουν παίξει κανένα ρόλο. Τίποτα δεν έγινε. Μετά από αυτά έχουμε την απόφαση ε, δημιουργίας ενός μηχανισμού ε, για την έρευνα των περιστατικών ε, στη μήκο της γραμμής επαφής το 2011 και το 2012 ο πρόεδρος Αρμενίας, ο πρόεδρος της Ρωσίας που ήταν ο Πούτιν και είναι ακόμα βέβαια και ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν αποφάσισαν να δημιουργήσουν αυτόν τον μηχανισμό στην διακήρυξη του Σότσε αλλά μόνο το Αζερβαϊτζάν άρχισε τη δουλειά σε αυτόν τον τομέα. Η ομάδα του Μίνσκ δεν έχει προχωρήσει. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Δεν, γίνεται, δεν κάνει τίποτα για την επιλύση του ζητήματος αυτού. Για μας λοιπόν για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σίγουρα έχει έρθει η ώρα να κάνουμε κάτι αν πιστεύουμε στην πολιτική γειτονία ε, και στην ειρήνη και στις διπλωματικές μας ικανότητε να ε, οδηγήσουμε άλλους λόγους στην ειρήνη. Και το ερώτημα μου προς είναι τι μορφή θα είχε ένας ε, ευρωπαϊκός μηχανισμός συμμετοχής. Γιατί όλο μιλάμε για αυτή την ανάγκη να συμμετάσχουμε, αλλά πώς θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε έναν τέτοιο μηχανισμό και πότε, διότι είναι απαραίτητη η παρουσία μας εκεί με νόμιμο τρόπο, με νόμιμη μορφή. Μπορούμε να κάνουμε όσες διακηρύξεις θέλουμε. Ότι μας αρέσει ο ένας ή ο άλλος, ε, ε, ότι υποστηρίζουμε τον ένα ή τον άλλο, αλλά δυστυχώς τελικά δεν κάνουμε τίποτα. Αυτά έχουν συμβεί εδώ και 20 χρόνια από τότε που ξεκίνησε αυτή η διαμάχη. Και τελευταία ερώτηση προς εσάς ε, στην τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση. Ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το επόμενο βήμα της Ρωσίας στην περιοχή, γιατί είδαμε τι έγινε στη Φωσετία, είδα ότι και στη Γεωργία υπάρχει ένα πρόβλημα. Τι θα γίνει με την υπερθυνιστερία. Ε, συνδέονται μεταξύ τους αυτές οι τρεις ε, διαμάχες. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να, να προσθέσω τη φωνή μου. Θα ήθελα να αναφερθώ στο ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει μια ταχεία αντίδραση της υποεπιτροπής μας. Είχαμε πρόσφατα, διαβάσει όλοι, τις πληροφορίες και τις αναλύσεις σε σχέση με αυτή τη σύγκρουση. Πρέπει να ομολογήσω τώρα ότι μετά από όλα αυτά τα οποία διάβασα και έμαθα, έχω τρία σχόλια. Πρώτα απ' όλα, οι κύριοι εμπλεκόμενοι σε αυτήν την ε, ε, διαμάχη είναι πάντα η ίδια η Ρωσία και η Τουρκία. Πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι έχουμε ορισμένα νέα στοιχεία στην συγκεκριμένη κατάσταση που έχουμε σήμερα ενώπιόν μας. Πρώτα απ' όλα, οι ίδια, ε, αντίμαχες χώρες, ιδίω το Αζερβαϊτζάν, περνάνε μια περίοδο, περίοδο οικονομικών δυσκολιών, αυξημένων οικονομικών δυσκολιών. Γι' αυτό βλέπουμε ότι υπάρχει η δυσφορία του πληθυσμού στις χώρες αυτές που είναι όλο και μεγαλύτερη. Ο πληθυσμός διαμαρτύρεται κατά της στάσεις της εξουσίας της χώρες αυτές. Και αυτή τη φορά η εντύπωση μου είναι ότι μέχρι κάποια τουλάχιστον χρονική στιγμή η κατάσταση που δημιουργήθηκε ήταν προς το όφελος και των δύο χωρών. Επίσης, να σταθούμε στη στρατιωτική πτυχή. Εγώ ανησυχώ ιδιαίτερα από το γεγονός ότι Κάθε φορά έχουμε τέτοιες ε, διαμάχες και αντιπαραθέσεις που μας καταδεικνύει ότι οι αντιμεχόμενες πλευρές έχουν όλο και πιο προωθημένο και βαρύ εξοπλισμό. Βλέπουμε να έχουν άρματα μάχης, να έχουν πυράβλους μεγάλου βεληνικούς. Βλέπουμε λοιπόν να υπάρχει μια κλιμάκωση σε ό,τι αφορά τη συγκέντρωση βαρέως οπλισμού σε αυτήν την περιοχή και αυτό φυσικά είναι κάτι το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο. Και τώρα να θέσω και δύο ερωτήματα στους καλεσμένους μας. Πρώτα απ' όλα, τι πιστεύετε σε σχέση με τη δυνατότητα να υπάρξει διεύνηση αυτής της ε, σύγκρουσης. πως το παρόν αυτή η σύγκρουση είναι γεωγραφικά περιορισμένη σε μια συγκεκριμένη περιοχή μονάχα αλλά έχουμε γύρω από την εστία της κρίσης και άλλες χώρες οι οποίες βρίσκονται σε διαμάχη μεταξύ τους. Υπάρχει ένας πραγματικός κίνδυνος αυτή η διαμάχη να διευρυνθεί και να περιλάβει και άλλες χώρες. Δεύτερο ερώτημα και το οποίο έχει να κάνει με την αδυναμία δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν βλέπουμε τις διάφορες ε, αναλύσεις για την κατάσταση αυτή. Βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όλο και περισσότερο κάνει βήματα προς το απίσω σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, σε ό,τι αφορά την ηγετική της στάση σε παγκόσμιο επίπεδο. Και εδώ θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά που είπε η κυρία Μανταπόλ. Θα θέλαμε να μας δώσετε και κάποιες ιδέες, κάποιες συστάσεις για το τι μπορούμε να κάνουμε. Τι μπορεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο μπορεί πάντα να συζητά, μπορεί να καταλήγει σε ψηφίσματα κτλ. Αλλά αυτά έχουν μικρή μοναχα επίπτωση στην κατάσταση επιτοπίως. Τι προτείνετε να κάνουμε λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ λέει και η πρόεδρος. Έχουμε ακούσει... Φτάσαμε στο τέλος του καταλόγου των ομιλητών. Ε, θα ήθελα λοιπόν τώρα και εγώ να πω δύο λόγια για τις παρεμβάσεις Πασκού και Τζέμκα και να μιλήσω για το ευρύτερο πεδίο εδώ και τους βασικούς εμπλεκόμενους. Βεβαίως ε, υπάρχει ανάγκη, όπως είπαν πολλοί, για μεγαλύτερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν και πιστεύω ότι η ανάγκη είναι ακόμα μεγαλύτερη. Ε, γιατί εδώ μιλάμε για αδράνεια του δυτικού κόσμου σε πολλές περιοχές συγκρούσεων. Αν δούμε αυτές τις σύντομες δηλώσεις ότι δηλαδή υπάρχει αποχώρηση των Αμερικανών λόγω των εκλογών. Δεν το πολύ πιστεύω αυτό. Οι αμερικανικές πολιτικές είναι πολύ πιο σταθερές. Η αμερικανική γερουσία είναι υπεύθυνη για θέματα εξωτερικής πολιτικής, ε, είναι βαθύς γνώστες όλων αυτών των θεμάτων. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε και αυτή τη διάσταση. Η κυρία Πόλα αναφέρθηκε στους Αμερικανούς. Θα πρέπει να δούμε μια ευρύτερη δυνατότητα δράσης της ομάδας του Μίνσκ. Ε, σίγουρα είναι ανάγκη να δράσουμε ταχύτερα Ίσως πρέπει να γίνει μια αναδιαμόρφωση της ομάδας του Μίνσκ. Γιατί υπάρχει ανάγκη ε, γρήγορων διαπραγματεύσεων και διαβουλεύσεων μεταξύ των ε, βασικών εμπλεκομένων. Για το Ιράν επίσης θέλω να ρωτήσω και εγώ κάτι όπως και οι προηγούμενοι. Είναι σημαντικός παίκτη Υπάρχει μεγάλη κοινότητα Αζέρων που βρίσκεται σε περιοχή του Ιράν, στο έδαφος του Ιράν και η πολιτική του Αζερμπαϊτζάν προς το Ιράν ήταν πάντα κάπως ιδιαίτερη διότι έπρεπε να λαμβάνει υπόψη και την ευημερία αυτής της κοινότητας και άρα υπήρχε διάλογος πέρα από τα πολιτικά γεγονότα. Υπάρχει λοιπόν δυνατότητα να ε, διευρύνω με το πεδίο δράση που είναι τώρα λίγο περιορισμένο και τους εμπλεκομένους. Επίσης, πώς βλέπετε στον ρόλο των πρόσφατων στρατιωτικών συμφωνιών. Α, πρόσφατον, όχι πρόσφατον, ναι, είναι κάποια χρόνια που συνήθισαν, αλλά είχα, ε, τροποποιήθηκαν πρόσφατα μεταξύ Ρωσίας και Αρμενίας. Αυτή η συμφωνία είναι ευρύτερη και έχει σχέση με την φιλοδοξία της Ρωσίας να ανακτήσει επιρροή σε πρώην σοβιετικά εδάφη, τα εδάφη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και να διασφαλίσει τη δυνατότητα ε, προστασίας και των παλαιών εδαφών της. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για πολλούς από εμάς. Μια τέτοια αντίληψη είναι πολύ επικίνδυνη. Θέλω λοιπόν να μου πείτε κι εσείς πώς βλέπετε αυτό το θέμα. Ε, λοιπόν, πρώτα θα μιλήσει η κυρία Μάντα Πολ που πρέπει να φύγει και μετά ο κύριος ε, Κιμάρες. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολλές οι ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω τις περισσότερες, ε, αλλά σύντομα. Πρώτα απ' όλα, το ζήτημα της οικονομίας του Αζερμπαϊτζάν. Δεν πρέπει να πιστεύουμε ότι η κλιμακούσα αυτή δεν θα είχε λάβει χώρα αν η αγορά δεν είχε καταρρεύσει και πήγαινε πολύ καλά οικονομικά το Αζερβαϊτζάν. Αυτό είναι κοντόφθαλμο ω άποψη. Όπως είπα στα σχόλιά μου, οι κλιμακώσει αυτέ εντείνονται τα τελευταία χρόνια, ε, ακόμη και σε εποχές που η οικονομία του Αζερβαϊτζάν πήγαινε εξαιρετικά καλά. Οπότε δεν πρέπει να έχουμε τη στενόμυαλη άποψη ότι η κατάρρευση της οικονομίας έπαιξε ρόλο. Για το ποιο υποφελείται από την διαμάχη είναι σαφέ. Τα μέρη που υποστηρίζουν το status τα μέρη που ε, εποφελούνται της για να συγκεντρώσουν τους πληθυσμού υπό μια εθνικιστική ιδεολογία και να του κάνουν να ξεχάσουν κάποια εγχωρία ζητήματα και φυσικά οι Ρώσοι οι οποίοι εκμεταλλεύονται τη διαμάχη για να ενισχύσουν τη δική του σχέση ανάμεσα στι δύο χώρε και ευρύτερα στην περιοχή. Νομίζω ότι αυτό είναι σαφέ. Θύματα όλων αυτών είναι οι πολίτε τη Αρμενία και του Αζερβαϊτζάν φυσικά. Συμπεριλαμβανομένων φυσικά όσων όλοι, όσοι έχουν μετατοπιστεί εσωτερικά μιλάμε για σχεδόν ένα εκατομμύριο ανθρώπου τα τελευταία 20 χρόνια παραμένουν χωρί. Ε, ε, σπίτι. Ε, ακόμα περιμένουν να γυρίσουν στα σπίτια του. Είναι μια θλιβερή ιστορία. Τώρα για το ρόλο τη Γεωργία. Η Γεωργία δεν παίζει ε, απευθεία ρόλο στην διαμάχη. Αλλά αν η διαμάχη αυτή κλιμακωθεί σημαντικά, θα έχει συνέπειε και για τη Γεωργία. Διότι είναι γείτονα χώρο. Οπότε η Γεωργία θα θέλει να επιληθεί η σύγκρουση αυτή το συντομότερο δυνατόν και με τρόπο που να μην συμπεριλαμβάνεται η ρωσική παρουσία τόπου. Γιατί αν υπάρχει ρωσική παρουσία ή κάποια ρωσική συμφωνία, αυτό θα ρηψοκινδυνεύσει ε, την όλη η περιοχή του Νοτιού Καυκάσου να πέσει ξανά υπό την ρωσική επιρροή. Αν επιτρέπετε να πω κάτι τέτοιο σήμερα. Τώρα για το ζήτημα του Ιράν για λόγους ασφαλείας ε, το Ιράν ε, φυσικά δείχνει κάποιο ενδιαφέρον αλλά αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα του είναι κάτι άλλο είναι η Μέση Ανατολή είναι η μάχη κατά του Ισλαμικού κράτους και το μέλλον της Συρίας αλλά φυσικά ε, ανισχύει το Ιράν για την διαμάχη αυτή και έχει δείξει κάποιες ε, ενδείξεις ότι θα ήθελε να συμμετάσχει σε κάποια ειρηνευτική διαδικασία ή να βοηθήσει να ξεκινήσει ένα ειρηνευτικό σχέδιο, αλλά έχει πει ελάχιστα στα μέσα. Η σχέση του Αζερμπαϊτζάν με το Ιράν δεν είναι μυστικό. Για πολλά χρόνια οι σχέσεις μεταξύ τους ήταν δύσκολες. Είχαν ακουστεί διάφορες ε, θεωρίες συνωμοσία μεταξύ των δύο για το ποιος κάνει τι αλλά πιστεύω ότι μετά από την αλλαγή ηγεσία στο Ιράν ε, με τον πρόεδρο Ρουχάνη ε, έχει αλλάξει το, η ατμόσφαιρα των σχέσεων μεταξύ τους ε, έγιναν πολλές διπλωματικές επαφές μεταξύ των δύο χωρών όλα ένα αυξάνεται τη συνεργασία, το εμπόριο, η ενέργεια οι μεταφορές υπάρχουν νέα έργα για διάφορους ε, οδούς μεταφορών. Οπότε ε, οι εποχές που το Ιρακ και το Αζερβαϊτζάν ε, είχαν μια πολύ δύσκολη σχέση μεταξύ τους έχουν παρέλθει και κινούμαστε προς μια πιο θετική, δυναμική σχέση. Κάτι καλό και για τις δύο χώρες και υποφέλες για την περιοχή και φυσικά και για την εξωτερική πολιτική του Αζερμπαϊτζάν αυτό είναι καλό διότι προσφέρει το Ιράν ένα αντιστάθμισμα σχέση με την παρουσία της Ρωσίας. Οπότε ε, είναι κάτι αισιόδοξο. Όσον αφορά την Τουρκία, δεν νομίζω ότι η Τουρκία μπορεί να κατηγορηθεί απευθεία για την πρόσφατη κλιμάκωση. Δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα ήταν δίκαιο. Δεδομένου αυτού όμως κάποια από τα σχόλια της τουρκικής ηγεσία όπου υποστηρίζουν τη μία μόνο πλευρά πιστεύω ότι θα μπορούσαν να είχαν γίνει λίγο πιο διακριτικά. Αλλά σαφώ η σχέση μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Τουρκία ε, έχει κάτι το ιδιαίτερο. Ε, λέμε συχνά δύο χώρε, ένα λαό, αλλά εγώ δεν συμφωνώ απαραίτητα με μια τέτοια δήλωση. Αλλά ξέρετε, υπάρχει και κάποια ιστορία σε όλο αυτό. Έχουν κάποιου στενού ε, στενέ ε, πολιτικέ σχέσει και οικονομικέ σχέσει. Το Αζερμπαϊτζάν είναι μεγάλο επενδυτή στην Τουρκία σε ενεργειακέ υποδομέ αυτή την εποχή. Συνεπώς είναι μια... Ε, έτσι η Τουρκία δεν μπορεί να συμμετάσχει ενεργά στη διαμάχη αυτή του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Δεν ξέρω κατά πόσο οι πολιτικέ του Ερντογάν τη σήμερα ημέρα είναι καλέ για την περιοχή. Η σημερινή εξωτερική πολιτική τη Τουρκία ε, οξύνει την ασφάλεια στην περιοχή αντί να βοηθά στην πρόθεση της Ειρηνή. Όλοι το γνωρίζουμε αυτό το Η Τουρκία κινείται προς ε, ε, ένα καθεστώς αρκετά αυταρχικό χωρίς ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα. Και αυτό θα οξύνει τη σχέση με τους ε, γείτονες χώρε. Όσον αφορά τη Ρωσία και την Αρμενία, πιστεύω ότι οι σχέσεις μεταξύ Ρωσία και Αρμενίας υπονομεύουν την ασφαλεία τη Αρμενίας. Είτε μιλάμε για τη στρατιωτική συμφωνία με την Αρμενία, είτε για τη σχέση της ε, ε, στην Ευρασιατική Ένωση. Όλα αυτά έχουν υποσκάψει την εθνική κυριαρχία της Αρμενίας και έχουν περιορίσει τις επιλογές που μπορεί να κάνει εσωτερικά και στην εξωτερική της πολιτική. Αυτό είναι σαφές για όλους. Οπότε έτσι η Αρμενία παραμένει βάλωτη. Και αυτό εξηγεί κάτι που έχουμε δει ήδη, ότι οι Άρμενοι έχουν οφηθεί λίγο να υποστηρίξουν μια ειρηνευτική διαδικασία της Ρωσίας επί τόπου. Κάτι που μπορεί να υπονομεύσει την κατάσταση. Τώρα για το ποιο ε, θα είναι φτιάξει ειρήνη και ποιο θα είναι φτιάξει πόλεμο στην περιοχή όσον αφορά τη Ρωσία, όλοι το γνωρίζουμε. Αυτό που είπατε είναι σωστό. Η δράση τη Ρωσία πρόσφατα στην Ουκρανία απέδειξαν ότι δεν επιθυμεί την ειρήνη, ότι βοηθά να κλιμακώνονται οι ε, διαμάχες ε, και να παγιώνονται οι διαμάχες ε, και η επίλυση αυτών των διαμαχών βασίζεται στους στόχους της Ρωσίας το οράμα της Ρωσίας στην εξυπηρέτηση του οράματος για το μέλλον της Ρωσίας πιστεύω ότι υπάρχει κίνδυνος να επεκταθεί η διανεξή αν κλιμακωθεί έχουμε καταφέρει να την περιορίσουμε μέχρι στιγμής αλλά δεν πρέπει να θεωρούμε αυτό τον περιορισμό δεδομένο Μπορεί να επεκταθεί αυτή η διαμάχη αν αρχίσουν να συμμετέχουν και άλλοι, άλλες χώρες της περιοχής. Κάτι που θα δυσχέρανε την κατάσταση. Σαν αφορά των ΗΠΑ. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, δεν έχουν αποσύρθει από τον Νότιο αλλά σε τελική ανάλυση αποτελούν ελάχιστη μελιτέα δύναμη ε, στην περιοχή ε, όσον αφορά την επιρροή τη. Και αυτό είναι φυσιολογικό. Αν σκεφτεί κανεί τι έχουν να αντιμετωπίσουν οι Ηνωμένε Πολιτείε, ειδικότερα στην Μέση Ανατολή, το Ισλαμικό κράτο, την ε, τρομοκρατική απειλή, τα εσωτερικά ζητήματα που είναι τεράστια, το Καραμπάχ σε τελική ανάλυση ε, είναι άγνωστο για τους Αμερικανούς. Ε, με δυσκολία θα μπορούσε κανείς, ένας Αμερικανός να βρει στο χάρτη τον Νότιο Κάφκασο. Δεν αποτελεί λοιπόν πρώτη προτεραιότητα, αλλά φυσικά αν κλιμακωθεί θα αποτελέσει πρώτη προτεραιότητα και όπως είπαμε αυτό το τόξο αστάθειας από την Ανατολική Ουκρανία θα φτάσει μέχρι την Αφρική μόνο σε τέτοια, αν φτάσει μέχρι την Αφρική μόνο τότε θα αποτελέσει προτεραιότητα για την Αμερική ε, αλλά όπως είπα δεν φανταζόμαστε να έχουμε κάποια σημαντική συμμετοχή των ΗΠΑ στο εγγύς μέλλον όταν εκλεγεί ο νέος πρόεδρος ε, δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ούτε τι πολιτικές θα ακολουθήσει Ευχαριστώ. κύριο κύριος Γκυμαράης έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους βουλευτές για τα σχόλια και τις ερωτήσεις τους. Και όπως ε, είπα και στα αρχικά μου σχόλια, είπα ότι παρά την ε, αυτοσυγκράτηση με την οποία πρέπει να εκφραστώ, τόνισα που βρισκόμαστε σε σχέση με τη σημασία αυτής της ε, σύγκρουσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση τόνισε τις προσπάθειες που έκανε η ύπατη εκπρόσωπος για την αντιμετώπιση του θέματος αυτού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν εμπλέκεται, δεν υπάρχει θέμα αδράνειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν ε, φυσικά <clears throat> πολλοί λόγοι να συζητήσουμε το πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η στάση και η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή αυτή. Αλλά όλα αυτά τα οποία πράττουμε στα πλαίσια του συμπεφωνημένου διεθνούς σχήματος όπως έχει απαρτιστεί από τους συμπρόεδρους της ομάδας του Μίνσκ. Η συμμετοχή στο σχήμα αυτό εξαρτάται από τις αποφάσεις του ΑΣΕ. Δεν είναι ότι εμείς απλώς μπαίνουμε και παρεμβαίνουμε σε μια τέτοια διαμάχη και αποφασίζουμε το ρόλο το δικό μας. Αυτό είναι κάτι που καταρχήν πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή γιατί πρόκειται για μια σύγκρουση που σοβεί εδώ και πολλά χρόνια. Αυτή τη στιγμή το διεθνές σχήμα το οποίο έχει αποφασιστεί είναι οι δύο συμπρόεδροι της ομάδας του ΜΙΝΣ και οι προσπάθειές τους είναι οι προσπάθειες που πρέπει να υποστηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή είναι η προσπάθεια που καταβάλει μη φιδωμένη προσπαθειών και η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής. Επομένως, η δική μας ε, στάση διέπεται από την ανάγκη να δείξουμε μια υπομονή για την ε, αντιμετώπιση των εξελίξεων. Φυσικά όλα αυτά που είπα, είπατε για τους εξωτερικούς ε, εμπλεκόμενους, όχι τους άμεσα εμπλεκόμενους και μόνο, φυσικά όλα αυτά είναι έγκυρα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο λάβαμε από εσά και το οποίο σίγουρα και εγώ το υποστηρίζω. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι, κλείνουμε έτσι το σημείο αυτό της σημερινής διάταξης. Έχουμε στη συνέχεια ένα πολύ ενδιαφέρον επόμενο σημείο. Θέλω να ευχαριστήσω και τους ε, δύο ομιλητές μας και θέλω να σας ευχαριστήσω και σας για την παρουσία σας στην συζήτηση και σας ευχαριστώ λοιπόν και για την ε, βοήθεια που έκανε και το Προεδρείο και το, η Γραμματεία της Υποεπιτροπής. Τώρα δεν έχουμε ακόμα τους ομιλητές. Μάλλον δεν έχουμε δυνατότητα δεύτερου γύρου συζήτησης για το θέμα αυτό, αλλά θα επανέλθουμε ως ο το θέμα αυτό. Παρακαλώ παραμείνετε στην αίθουσα για το επόμενο σημείο. Καθίστε παρακαλώ κυρίες και κύριοι, να αρχίσουμε με το επόμενο θέμα μας, που είναι η καταπολέμηση του Ισλαμικού κράτους στις χώρες της Ανατολικής και της Νότιας Γειτονίας. Είναι μεγάλη μου χαρά να παρουσιάσω τους ε, δύο διακεκριμένους προσκεκλημένους μας, την κυρία Φλωράνς Γκάου, πανώτερη αναλήτρια στο Ινστιτούτο Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα ασφάλειας και τον καθηγήτρια, ο καθηγητή Ανάρ Βαλίγεφ, αντιπρόεδρα ακαδημαϊκών υποθέσεων στο Πανεπιστήμιο Αίντα του Μπακού. Νομίζω ότι υπάρχει κάποια συμφωνία σε σχέση με τον καταμερισμό εργασίας μεταξύ των δύο προσκεκλημένων μας. Η συζήτηση θα εστιάσει σε μια ευρύτερη περιοχή. Και σήμερα θα κάνουμε ευρείες διαβουλεύσεις. Το Ισλαμικό κράτος είναι παγκόσμια απειλή πολλά από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά αξιολογεί την κατάσταση και εξετάζει μέτρα πρόληψης και αποτροπής του Ισλαμικού κράτους και ε, του ρόλου του διεθνώς. Σίγουρα θα είναι ενδιαφέροντα αυτά που θα μας πούν οι δύο προσκεκλημένοι μας και μετά βεβαίως θα ήθελα να γίνει μια ωραία συζήτηση. Πρώτα θα κάνει την παρουσίασή της η κυρία Φλωράνς Γκάουπ και μετά ο καθηγητής Άναρ Βαλίεφ. Μετά θα γίνει συζήτηση με ερωτήσεις, απαντήσεις. Και αν μπορέσουμε θα έχουμε και ένα δεύτερο γύρο ερωτήσεων απαντήσεων. Η κυρία Γκάουμπ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ που με ξαναπροσκαλέσατε. Στα λίγα λεπτά που έχω στη διάθεσή μου θα ήθελα να κάνω τέσσερις στρατηγικές παρατηρήσεις όταν πρόκειται για τη μάχη κατά του ISIS, κυρίως στον Νότο. Πού βρισκόμαστε καταρχήν σε σχέση με τις εξελίξεις στον Νότο. Υπάρχει μια συμμαχία που 22 χωρών που ανέλαβε στρατιωτική δράση κάποια αριθμητικά στοιχεία. Περίπου 11.000 ε, ε, αεροπορικές επιδρομές έγιναν στην περιοχή, το 70% στο Ιράκ και το 30% στη Συρία. Οπότε η μεγάλη πλειοψηφία γίνεται στο Ιράκ των πληγμάτων. 33.000 στόχοι κατεστράφησαν. Ε, βεβαίως ε, υπήρχε και κάποια απώλεια εδάφους από την πλευρά του ISIS, αλλά γενικά η οργάνωση δρά επιθετικά αλλού. Ε, υπήρξαν κάποιες επιτυχίες στις μάχες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει ε, ακόμα ε, προοπτική στρατηγικής νίκης. Η, είναι υβριδική η μορφή του ISIS, μπορεί παράλληλα να είναι πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Ε, ε εδαφική, ε, εικονική, συμβατική, ασύμετρη, ε, δεν είναι μία, ε, δεν είναι ένα το πεδίο μάχης αλλά περισσότερα και περνώ τώρα σε ορισμένα στρατηγικά θέματα που θα ήθελα να σας παρουσιάσω. Το πρώτο είναι ότι ως Ευρωπαίοι τίνουμε να βλέπουμε ε, μέσα από το φακό της Συρίας το ISIS, γιατί είναι πιο κοντά η Συρία σε εμά, γιατί πολλοί Σύριοι ήρθαν στην Ευρώπη για να γλιτώσουν, αλλά το πρόβλημα δεν γεννήθηκε στη Συρία. Άρα δεν θα λυθεί και στη Συρία. Ένας λόγος, και τον αναφέρατε εσείς κυρία Πρόεδρε, είναι ότι 5.000 Ευρωπαίοι, όπως γνωρίζετε, έχουν ενταχθεί στο ISIS ή πέρασαν από εκεί και οι μισή περίπου γύρισαν πίσω στην, Ευρω... στην υπηρετική Ευρώπη. Οπότε, ανεξάρτητα από το τι θα γίνει στη Ράκα, οι άνθρωποι αυτοί έχουν έρθει εδώ και ενδεχομένως όχι όλοι, αλλά οι μισοί αποτελούν δυνητική απειλή. Υπάρχει σαφή σύνδεση μεταξύ της εμπειρίας που είχαμε στα εδάφη του ISIS και στις τρομοκρατικές δραστηριότητες. Δεν λέω ότι όλοι που θα γυρίσουν από τη Συρία είναι τρομοκράτες, αλλά ισχύει το αντίστροφο. Τα τρομοκρατικά πλήγματα που είδαμε την τελευταία τριετία αρχίζοντας στο, στις Βρυξέλλες στο Εβραϊκό Μουσείο, όλα έγιναν από ανθρώπους που γύρισαν από τη Συρία και το Ιράκ και αποτελούν σοβαρή πρόκληση για μας τους Ευρωπαίους. Ε, έχουν θολώσει γραμμές μεταξύ εξωτερικής πολιτικής και εσωτερικής πολιτικής ασφάλειας. Τα, οι πρώτοι που τώρα θα περάσουν ε, από δίκη στην Ευρώπη και επειδή διάπραξαν ε, εγκλήματα στη Συρία ή στο Ιράκ οι ποινές είναι 4 με 6 χρόνια, όχι παραπάνω. Αυτή λοιπόν είναι μια πρόκληση η οποία βρίσκεται εκτός δικών μου, δικής μου ειδικότητας, αφορά περισσότερο εσά από και εμένα, εγώ δουλεύω στην περιφέρεια. Αλλά αυτό δείχνει ότι υπάρχει σαφής ευρωπαϊκή διάσταση στο θέμα, που δεν θα σταματήσει όταν πέσει η ράκα. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο σημαντικό θέμα που πρέπει να σημειώσετε, ότι τα παιδεία μαχών είναι πολλά, δυστυχώς ένα πεδίο είναι η Ευρώπη και αυτό δεν αλλάζει. Γιατί οι 5.000 Ευρωπαίοι 2.500 μπορεί να γύρισαν, είναι Ευρωπαίοι στον τρόπο δράσης και σκέψης τους. Χρησιμοποιούν το χώρο ε, Σέγγεν, ε, ε, χρησιμοποιούν τις αδυναμίες μας για να επικοινωνήσουν, να ταξιδέψουν και να λειτουργήσουν μέσα στο χώρο μας. Έχουν εμπειρία μάχης από αλλού, αλλά ξέρουν την Ευρώπη και τα κίνητρά τους ε, είναι ευρωπαϊκά. Το ISIS είναι παγκόσμιο φαινόμενο, αλλά τα κίνητρα των Ευρωπαίων ε, για να μπουν στον ISIS είναι ευρωπαϊκά. Δεύτερον, το μπαλόνι, το οποίο άμα το πιέζεις ε, ε, αλλάζει σχήμα, αλλά δεν σκάζει κατά ανάγκη. Αν δούμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του ISIS σήμερα, βλέπουμε ότι υπερεκτιμούμε το τι μπορούν να επιτύχουν οι αεροπορικές ε, ε, επιδρομές. Το γεγονός ότι ε, πολλές φορές σκεφτόμαστε ότι αν έχουμε πολλά θύματα θα εκλείψει το πρόβλημα. Μετατίθεται αλλού όμως. Οι μαχητές δεν πέφτουν θύματα των αεροπορικών επιδρομών, πάνε αλλού. Και αν δούμε ότι το ISIS είναι συνέχεια ε, κινημάτων που άρχισαν το 80 στο Αφγανιστάν, βλέπετε ότι ε, μεταξύ των στελεχών τους υπάρχουν ε, παλιά, μπαρουτοκαπνισμένα θα λέγαμε, στελέχη που πήγαν στην Τσετσενία, στη Βοσνία, στο Ιράκ, στη Συρία. Και πού θα πάνε μετά. Εγώ υποθέτω ότι θα πάνε μάλλον στη Λιβύη ή και την Αίγυπτο στον Ήλο. Στην Λιβύη τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι τον τελευταίο χρόνο ε, το ISIS κατάφερε να διπλασιαστεί και να φτάσει σε 6.000 μαχητές. Δηλαδή, αν λάβουμε υπόψη μας ότι η Λιβύη, έχει 6 εκατομμύρια κατοίκους, μικρή χώρα σχετικά, έχει περισσότερους μαχητές από τη Συρία από ότι ε, ε, έχουμε εμείς ως Ευρωπαίοι. Αυτό είναι ανησυχητικό. Βλέπουμε λοιπόν μετατοπίσεις μετά τις αεροπορικές μεταδρομές, ε, επιδρομές, αυτό δεν σημαίνει ότι λύνεται το πρόβλημα. Πάνε αλλού οι μαχητές. Κάτι άλλο που με απασχολεί σε σχέση με το φαινόμενο του μπαλονιού είναι ότι αν δούμε τη Λιβύη σήμερα και τις διαπραγματεύσεις και την προσπάθεια εξέβρεσης πολιτικής λύσης, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει διάσταση της ασφάλειας στην πολιτική αυτή συμφωνία. Ακόμα και αν έχουμε πολιτική συνένεση, παρόλα αυτά δεν έχουμε δώσει απάντηση στον κατακαιρματισμένο χώρο της Λιβύης, ε, τους πολέμους ε, που πολεμούν ο ένας τον άλλον. Είναι κατακαιρματισμένο το θέμα της ασφάλειας στη Λιβύη. Άρα λοιπόν, αν βρεθεί πολιτική συμφωνία, δεν σημαίνει ότι θα λυθούν τα προβλήματα όπως είναι σήμερα στη Λιβύη. Τρίτον, το Ιράκ. Είπα και προηγουμένως ότι το ISIS το θεωρούμε ως φαινόμενο συριακό, αλλά ε, στις γραμμές του ISIS κυρίως είναι Ιρακινή, η μισή ε, είναι Ιρακινή, η ηγεσία είναι Ιρακινή 100% αν και ο διοικητής της ε, Συρίας ήταν Ιρακινός πριν πεθάνει. Ε, διέπεται από τους Ιρακινούς λοιπόν δεν το λέω για να τους κατηγορήσω το Ιράκ, αλλά πρέπει να καταλάβουμε το Ιρακινό πλαίσιο που είναι σημαντικό. Ε, είχαμε και άλλα κινήματα και αλλού βέβαια, αλλά εκεί που ενισχύθηκε είναι ε, στο Ιρακινό πλαίσιο μετά το 2003. Εκεί ενισχύθηκε το Ισλαμικό κράτος. Και θα πρέπει να υπογραμμίσουμε λοιπόν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στο Ιράκ, ούτως ώστε η σουνητική κοινότητα να ε, ενταχθεί πάλι στο πολιτικό παιχνίδι. Ο Πρωθυπουργό προσπαθεί σίγουρα πολύ σκληρά, αλλά δεν έχει τόση πολιτική υποστήριξη στο Κοινοβούλιο, το Ιρακινό Κοινοβούλιο, όπως θα θέλαμε. Ίσως ακούσατε τις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις αυτών των ημερών. Ιράκ λοιπόν, το Ιράκ είναι το πρώτο, είναι στην πρώτη γραμμή σε πολιτικό επίπεδο το Ιράκ όταν πρόκειται για την καταπολέμηση του ISIS στο Νότο. Η Συρία είναι μάλλον παρεπόμενο. Αν δούμε, αν λυθεί η σύγκρουση στη Συρία, δεν θα λυθεί το φαινόμενο του ISIS, γιατί προέκυψε, ε, ε, δεν γεννήθηκε εκεί, αλλά προέκυψε από άλλα προβλήματα. Εγώ νομίζω ότι επειδή γεννήθηκε στο Ιράκ, πρέπει το ISIS να πεθάνει και στο Ιράκ. Τέλος, ε, η τελευταία μου στρατηγική παρατήρηση είναι ότι δυστυχώς ενώ τα τελευταία πέντε χρόνια συζητούμε για το τι σημαίνει η Αραβική Άνοιξη που μπορεί να πάει, ε, η στρατολόγηση ε, συνεχιζόταν όλο αυτό το διάστημα. Το 2000, ε, από το 2011 η κατάσταση επιδεινώθηκε. Η ανεργία των νέων που ήταν 27 με 29% ανέβηκε κατά δύο μονάδες για διάφορους λόγους. Ε, γιατί λόγω θεμάτων ασφαλείας η οικονομία δεν μπορούσε να λειτουργήσει και πιο σημαντικό λόγω της δημογραφικής εξέλιξης στην περιοχή. Τα επόμενα 4-5 χρόνια λοιπόν η περιοχή θα πρέπει να δημιουργήσει 80 εκατομμύρια θέσεις εργασίας για να διατηρήσει την ανεργία των νέων στα σημερινά επίπεδα. Ε, αυτό Στι κοινωνικέ επιστήμες, όταν έχουμε ανεργία των νέων 30%, ε, έχουμε μεγάλο κίνδυνο πολιτικών ταραχών. Ως επιτοπλίστων, ε, δε, δεν έχουμε φτάσει στο ε, ανώτατο σημείο της ανεργίας. Το λέω αυτό γιατί είναι ε, ένα ανησυχητικό φαινόμενο σε όλες τις περιοχές. Και στην Τινησία που έχει στη Συρία στείλει 4-5 μαχητές αλλά και ε, την ε, Σαουδική Αραβία που έχει μεγάλη ανεργία. 3.000 ε, από τη Σαουδική Αραβία στο Ιράκ πήγαν στο ISIS. Οπότε και στο, στις χώρες του κόλπου η πρόκληση είναι μεγάλη. Ε, το σύστημα πρόνοιας δεν εγγυάται την πολιτική σταθερότητα. Επίσης, οι, οι ίδιοι λόγοι που δημιούργησαν πρόβλημα το 2011 εξακολουθούν να υφίστανται. Ε, Εμεί ε, θέλουμε να φτάσουμε στη συνεργασία της ασφάλειας πριν από το 2011, αλλά αυτό είναι δύσκολο διότι ε, αφού το ανέλαβε ο πρόεδρος ε, Σίση τα ε, πράγματα επιδεινώθηκαν. Ε, τριπλασιάστηκαν οι επιθέσεις από την ανάληψη της Προεδρίας. είναι πολιτικό εγχείρημα η καταπολέμηση των εξεγερμένων εμείς μπορούμε να το δούμε αυτό και από το Αφγανιστάν. οι εξηγέρσεις είναι πολιτική έκφραση ε, λειτουργούν κάποιε μονάδε του ISIS με αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό χρειάζεται πολιτική απάντηση. Δεν θέλω να πω ότι πρέπει να απευθυνθούμε στο σκληρό πυρήνα, αλλά κάθε εξέγερση περιβάλλεται από πληθυσμό, από κόσμο που του ε, βοηθάει. Μπορούμε να το δούμε στο Σινά, όπου υπάρχει, αυτός, ε, υπάρχει το, το, το τοξικός γάμος με του Βεδουίνου που δεν έχουν να κάνουν με το Ισλάμ, αλλά έχουν τα ίδια παράπονα απέναντι στο Κάιρο με το ISIS. Αυτή είναι η τελευταία μου παρατήρηση. Το ISIS είναι μια οντότητα πολύ βίαιη, αποτρόπαιη, αλλά τι προσφέρει πέρα από αυτά. Δίνει ε, προοπτική επαναστατική στους νέους που δεν έχουν άλλη εναλλακτική. Άρα λοιπόν οι χώρες εταίρημα στην περιοχή τι προσφέρουν. Πρέπει να προσφέρουν αλλαγή. Πρέπει να προσφέρουν ένα μήνυμα ελπίδας και επικοδομητικών εναλλακτικών, γιατί σε τελευταία ανάλυση είναι αυτή η επαναστατική χρειά που κάνει το ISIS ελκυστικό ε, στους νέους που δεν έχουν ε, να ελπίσουν σε τίποτα άλλο. Και σταματώ εδώ. Ευχαριστώ. Ήταν πάρα πολύ συναρπαστικά αυτά που μας είπατε. Καθηγητά κύριε Βαλίεφ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φωτίγα. Θέλω καταρχήν να σας ευχαριστήσω που μας προσκαλέσατε. Εδώ είναι μια μεγάλη τιμή και χαρά για μένα. Αυτό που θα προσπαθήσω να σας πω τα επόμενα δέκα χρόνια, 10 λεπτά συγγνώμη, είναι μια επισκόπηση για τους κινδύνους που επέχουν οι χώρες του Νότιου Καυκάσου για τον ευρωπαϊκό χώρο. Γιατί ακούτε πολλά στα μέσα ενημέρωσης για αυτούς οι οποίοι έρχονται από διάφορες περιοχές μαχητές του Ισλαμικού κράτους. Ο Νότιος Καύκασος είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση γιατί βρίσκεται στα σύνορα της Ευρώπης και το ερώτημα είναι κατά πόσο στο μέλλον αυτές οι περιοχές του Νοτιού Καυκάσου μπορούν να δημιουργήσουν ένα κίνδυνο για τον ευρωπαϊκό χώρο ως ε, χώρος ε, διέλευσης ή ως κέντρο τρομοκρατικών δραστηριοτήτων. Όταν μιλάμε για τον Νότιο Κάφκασο, μιλάμε περισσότερο για δύο χώρες, Γεωργία και Αζερμπάιτζαν. Η Αρμενία είναι μια μόνο εθνοτική χώρα με ομοιογενή πληθυσμό, αντίθετα από την ε, Γεωργία και το Αζερμπαϊζάν, που παρά τον ε, κοσμικό χαρακτήρα του κράτους θεωρείται παραδοσιακά ως μια μουσουλμανική χώρα. Και 75% του πληθυσμού του Αζερμπαϊτζάν είναι Σιήτες και μόνο 25% είναι Σουνίτες, ενώ στη Γεωργία περίπου 10% είναι μουσουλμάνοι, θεωρούνται μουσουλμάνοι, Πολλοί από αυτούς είναι εθνοτικά Αζεροί, είναι από την Τσετσενία ή από τον Ταϊστάν και από αυτό το 10% περίπου το 1 τρίτο είναι μάλλον 20% είναι Σίτες ε, και τα 80% είναι Σουνίτες. Τι έγινε λοιπόν μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, γιατί και οι δύο χώρες ήταν κομμάτια της Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε είχαν ζήσει σε απομόνωση από τον υπόλοιπο μουσουλμανικό κόσμο. Μετά από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης άρχισε να ξεκινάει μια προσπάθεια δίσδυσης διαφόρων Ισλαμικών ιδεολογιών. Η αλλαγή αυτή στην κοινωνία οδήγησε σε πολλά θετικά αποτελέσματα αλλά και πολλά αρνητικά αποτελέσματα. Αυτή η χώρα λοιπόν είναι και ένα κέντρο αστάθειας γιατί από τη μία πλευρά είναι το Ιράν, από την άλλη πλευρά η Τουρκία, ε, στα, στα βόρεια είναι ο Κάφκασος και υπάρχουν ε, το, το Νταϊεστάν, η Οσετία, η Καρμαναρία, περιοχές που έχουν πολύ μεγάλη δημογραφική αύξηση. Επομένως, η, υπάρχει αυτή η δημογραφική αύξηση στην περιοχή, αλλά δεν αντιπροσωπεύει κάτι το ιδιαίτερο για το Ισλαμικό κράτος αυτή η περιοχή, κυρίως στο Αζερμπαϊτζάν, Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού είναι Σιήτες και στην ε, Γεωργία είναι μη μουσουλμάνοι, κοσμικού χαρακτήρα μουσουλμάνοι. Στην δεκαετία του 1990, στο τέλος, οι σαλαφιστικές ομάδες δίδυσαν στο Αζερβαϊτζάν και στην Γεωργία αλλά δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλος ο αριθμός αυτών που ήταν ε, ε, προσκύμενοι στα σαλαφιστικά ρεύματα κάτω από 10.000 και όχι ιδιαίτερα ριζοσπαστικοποιημένοι. δεν είχε λοιπόν μεγάλο ενδιαφέρον για το Ισλαμικό κράτος αυτή η περιοχή. Σήμερα το Ισλαμικό κράτος συνστατολογεί ε, ανθρώπου για να πολεμήσουν τη Συρία από διάφορε περιοχέ, Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική, αλλά και μία από τι πιο ενδιαφέρουσε περιοχέ για προσιλητισμό μαχητών είναι η Ρωσία και οι πρώην δημοκρατίες της ε, Σοβιετικής Ένωσης. Οι, περιοχές λοιπόν αυτές του Καυκάσου είναι ένα πολύ ενδιαφέρον τοπίο για στρατολόγηση μαχητών. Όπως και στη Μέση Ανατολή, οι δημοκρατίε αυτέ έχουν τεράστια προβλήματα ανεργία, ανεργία των νέων, υπάρχει δυσφορία των νέων που θεωρούν ότι έχουν αποκλειστεί από το πολιτικό γίγνεσθε και πάρα πολλοί δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Ιδίω οι νέοι και δημογραφικά αυτέ οι περιοχέ έχουν μεγάλη αύξηση του πληθυσμού. Οι περισσότεροι νέοι λοιπόν είναι άνεργοι, βρίσκουν ιδιαίτερα ελκυστικέ τι ιδέε του Ισλαμικού κράτου. Από αυτή την άποψη, αν δείτε το χάρτη, η περιοχή του Βορρά, του Καυκάσου, το Ταταρστάν Παγκοσχά, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περιοχή για να μπουν στο Ισλαμικό κράτος. Υπάρχουν οι δυνατότητες να πετάξουν κατευθείαν μέσα από το Αζερβαϊτζάν και μετά μέσα από το Αζερβαϊτζάν να πάνε στην Τουρκία και από την Τουρκία στη Συρία ή μπορούν να πάνε πάλι στο Αζερβαϊτζάν, στη Γεωργία και να κατέβουν στην Συρία και το Ιράκ. Είναι εύκολη λοιπόν η μετάβασή τους χωρίς να κινήσουν υποψίες. Η περιοχή λοιπόν αυτή δεν είναι κέντρο ε, στρατολόγησης, είναι κυρίως κέντρο διέλευσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτές οι χώρες δεν έχουν και μαχητές που έχουν πολεμήσει στη Συρία. Υπάρχουν μαχητές από την Γεωργία και το Αζερμπαϊτζάν που είναι τώρα στη Συρία και στο Ιράκ. Βέβαια δεν ξεπερνάνε τους 250-300 ανθρώπους που είναι οι μαχητές του Ισλαμικού κράτους. 250 ίσως 300 από το Αζερβαϊτζάν, το πολύ 100 από την Γεωργία ή από την ε, Τσετσενία που βρίσκονται στη Συρία. Πολλές φορές κάνουμε το λάθος να πιστεύουμε ότι αυτοί που πολεμούν στη Συρία πολεμούν όλοι μέσα στα πλαίσια του Ισλαμικού κράτους. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Υπάρχει μια σημαντική μειονότητα αζερή που πολεμούν με την ομάδα Τζαμπάτα Αλ-Ρούσρα. Γιατί στην αρχή όταν πήγαν οι περισσότεροι εκεί, οι δύο φορέ αυτοί ήταν ενωμένοι, δεν είχαν ακόμα διασπαστεί. Οι περισσότεροι λοιπόν πήγαν σε αυτού το φορέα και πολλέ φορέ πολεμούσαν και με του Γεωργιανού μαζί με την ομάδα του Αμπούμα Ασοστανή, ο οποίο ε, είναι από την Γεωργία στην πραγματικότητα, ήταν πολεμιστής κατά της Ρωσίας στον πόλεμο της Γεωργίας, αλλά κατέληξε στη Συρία και ε, ο Μπατρινασβίλη, ο οποίος υποτίθεται ότι σκοτώθηκε το 2016 και ήταν ε, μαχητής λοιπόν του Ισλαμικού κράτους. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί Γεωργιανοί οι οποίοι προέρχονται από αυτή την περιοχή και οι οποίοι βρίσκονται στη δύναμη αυτή και στην ε, δύναμη της Τζαμπάτα Αν κοιτάξουμε λοιπόν τις στατιστικές για τους <clears throat> προερχόμενους από αυτή την περιοχή, βλέπουμε ότι είναι οριακός ο πληθυσμός των μαχητών από τον Κάφκασο. Ακόμα και οι 250 ή η μισή από τους 250 αν γυρίσουν στο Αζερμπάιτζαν αποτελούν ένα δυνητικό κίνδυνο. Θέλουν να γυρίσουν όμως οι περισσότεροι που πήγαν στη Συρία πήγανε στη Συρία με την οικογένειά τους. Δεν θέλουν να ξαναγυρίσουν γιατί η ιδεολογία τους τους ε, λέει ότι έκαναν ένα είδος εγύρας, έκαναν μια μετάβαση από την διεφθαρμένη κοινωνία της πατρίδας τους και πήγανε να ε, μιμηθούν το παράδειγμα του προφητή Μωάμετ όταν πήγε από την ε, από τη Μεδίνα στην, ε, στη Μέκα. Φύγανε λοιπόν από το διεφθαρμένο καθεστώς για να ζήσουν σε ένα καθαρό χαλιφάτο. Δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουν λοιπόν στις χώρες τους. Και τι θα γίνει αν καταστραφεί το Ισλαμικό κράτος κάτι το οποίο θα γίνει ίσως κάποια στιγμή. Πάλι αυτοί δεν θα γυρίσουν στην περιοχή του Βορειού Καυκάσου, του Νότιου Καυκάσου. Θα πάνε, όπως είπε η συναδελφός μου, είτε στο Ιράκ, είτε στην Αίγυπτο ή κατά πάσα στη Λιβύη. Ακόμα όμως και σε αυτήν την περίπτωση είναι δύσκολο να μιλήσουμε για μια εποχή μετά το Ισλαμικό κράτος. Τι θα γίνει να κατασταθεί δηλαδή το Ισλαμικό κράτος. Υπάρχει κίνδυνος που προέρχεται από αυτούς τους ανθρώπους ή όχι. Εγώ και πάλι πιστεύω ότι δεν είναι πολύ πιθανό αυτοί οι άνθρωποι να συνεχίσουν να κάνουν τρομοκρατικές ενέργειες ακόμα και αν γυρίσουν. Το σύστημα ασφαλείας του Αρσεμπαϊζάν είναι ιδιαίτερα σκληροτράχυλο και οι περισσότεροι από αυτούς που γυρίζουν από την Συρία περνάνε ανακρίσεις και πολλές φορές οι περισσότεροι φυλακίζονται είτε αποτελεί παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν έχει σημασία. Αυτό όμω είναι η πολιτική τη κυβέρνηση του Αζερβαϊτζάν τα τελευταία δέκα χρόνια. Με απλοϊκό τρόπο, οποιοδήποτε έρχεται από τη Συρία σημαίνει για αυτού ότι έχει πολεμήσει εκεί. Αν έχει πολεμήσει, είναι ποινικό αδίκημα, έχετε συμμετάσχει σε κάποια ομάδα μισθοφόρων, στη στενή κατευθείαν. Έτσι λοιπόν, πολλά άτομα που, ήταν, που έχουν γυρίσει από το Αζερβαϊτζάν έχουν μπει στη φυλακή, 14 με 16 χρόνια φυλακής κατά μέσον όρο. Θα υπάρξει λοιπόν απειλή από το Αζερβαϊτζάν και την περιοχή του Νοτιού Καυκάσου ως κέντρο στρατολόγησης ε, μαχητών. Θα είναι κίνδυνος για την Ευρώπη. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι απίθανο. Εγώ δεν πιστεύω μπορούν να υπάρξουν μεγάλες ομάδες τρομοκρατών που θα έρθουν στην Ευρώπη για να κάνουν τρομοκρατικές ενέργειες. Οι περισσότεροι από αυτούς αν δείτε ποιο στρατολογεί το Ισλαμικό κράτο και ποιου θέλει στην Ευρώπη, αυτοί που έρχονται στην Ευρώπη είναι προφανώ οι Ευρωπαίοι που μιλά θαυμάσια αγγλικά, φλαμανδικά, γαλλικά ή οτιδήποτε τέτοιο. Οι Γεωργιανοί και οι Αζερβαϊτζανοί δεν έχουν αυτέ τι γλωσσικέ γνώσει, δεν έχουν τη δυνατότητα να κυκλοφορούν ελεύθερα στον ευρωπαϊκό χώρο γιατί έχουν και περιορισμού σε σχέση με τις προξενικές θεωρίες κτλ. Τι μπορεί να κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει αυτή την περιοχή. Σας λέω και πάλι, ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διέλευσης και το Αζερμπαϊτζάν και η Γεωργία είναι ελκυστικοί χώροι για το Ισλαμικό κράτος, μόνο ως χώροι διέλευσης. Αν οι δυνάμεις ασφαλείας των δύο αυτών χωρών μπορέσουν να σταματήσουν τη διέλευση αυτών των ανθρώπων από τα σύνορα, αυτών που έρχονται από το Βόρειο Κάφκασο ή από την Ρωσία, αυτό θα είναι πραγματικά ένα σημαντικό πλήγμα προς το Ισλαμικό κράτος. Αυτά λοιπόν ήθελα να σας πω και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ενδεχόμενα ερωτήματα. Ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστήσω και τα δύο μέλη του πάνελ για αυτό τον πρώτο γύρο και ξεκινάει η συζήτηση. Ο πρώτος ε, ε, Φρόιντ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ για αυτούς τους εξαίρετους προσκεκλημένους που βρίσκονται ξανά εδώ. Η κυρία Γκάουμπ βρισκόταν εδώ πριν από 1,5 χρόνο νομίζω. Και αυτό με οδηγεί στην πρώτη μου παρατήρηση. Δυστυχώς ε, δεν ε, έχω κρατήσει σημειώσεις όπως κάνω συνήθως. Ε, θα ήθελα να δούμε βάσει το σημείο που είχα κρατήσει την τελευταία φορά που ήσασταν εδώ, αν όντω ίσχυσαν αυτά ε, βάσει, τον εξελι... του πώ εξελίχθηκε το ISIS. Ε, οπότε, εσεί τώρα θα πρέπει να θυμηθείτε αν κάποια από τα πράγματα που είχατε προβλέψει τότε τελικά έγιναν διαφορετικά. Ωστόσο, ακούγεται ένα επιχείρημα και εγώ δεν είμαι εμπειρογνώμων για να το αποδείξω σωστό ή λάθο, ότι η ψυχολογία παίζει σημαντικό ρόλο στην στρατολόγηση των αλλοδαπών μαχητών. Σύμφωνα με το επιχείρημα αυτό, είναι ευκολότερο να βρει κανεί ε, να στρατολογήσει μαχητέ όταν είναι επιτυχή, όταν επιτυχάνει του στόχου του. αλλά οι απώλειες ε, στο πεδίο μάχης ε, όταν αυτές γίνονται ε, εντονότερες τότε χάνει κανείς οπαδούς και οι οπαδοί απογοητεύονται. Θέλω να μου πείτε την άποψή σας γι' αυτό. Και δεύτερον, είπατε για ένα άλλο θέμα όσον αφορά τη Λιβύη. Είπατε ότι, δεν το βρίσκω τώρα, είπατε κάτι ότι Ε, οποιαδήποτε πολιτική συμφωνία στη Λιβύη δεν θα συνεπάγεται κάποια ασφάλεια. Και αναρωτιέμαι, η όλη διαπραγματευτική διαδικασία που λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή στη Λιβύη και που καθοδηγείται από αυτό το ζήτημα της ασφάλειας ε, ε, γιατί τι γίνεται εκεί πέρα από το κόμπλε υπάρχει το ζήτημα ασφαλείας που χαρακτηρίζει όλες του τις δράσεις. Γι' αυτό τον λόγο θέλει να πει και στα δύο μέρη εκεί να ε, συνέλθουν κάπως γιατί και αυτοί τους λέει, και εσείς τους λέει θα αποτελέσετε θύμα αυτής της έλλειψης ασφάλειας οπότε αυτό ήθελα να σας ρωτήσω ευχαριστώ ευχαριστούμε πολύ κυρία Νικολάη για άλλη φορά ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε να σας ε, ξανασυγχαρώ για τους προσκεκλημένους που επιλέξατε για αυτή τη συζήτηση να ευχαριστήσω και τους δύο μιλητές για τις παρεμβάσεις τους. Όταν ξεκίνησε η Αραβική Άνοιξη, ξεχάσαμε ότι οι τέσσερις εποχές του Βιβαλντή είναι τέσσερις εποχές. Ξεχάσαμε λοιπόν τις άλλες τρεις εποχές. Έχουμε ξεχάσει το χειμώνα και τώρα έχουμε κάποιο είδους αραβικό χειμώνα, ο οποίος ελπίζω να παραμείνει αραβικός και να μην επεκταθεί σε άλλες περιοχές. Συμφωνώ με την κυρία Φλόρανς Γκάουμπ όταν λέει ότι το έρχεται από το Ιράκ, έρχεται και από το Αφγανιστάν. Ξέρετε, οι πρώτες του ρίζες ε, έρχονται από το Αφγανιστάν. Ε, εκεί είχαμε τους αδερφούς μουσουλμάνους, και... αλλά το Ιράκ ήταν εκείνο που από το μέρος από όπου ξεκίνησε αυτό το φαινόμενο γιατί μιλάμε για φαινόμενο, δεν πρόκειται για κράτος. Είναι ένα ενδιαφέρον φαινόμενο, ε, δύσκολο στην αντιμετώπιση. Έχει μία πολιτική και μία ιδεολογική συνιστόσα που είναι πιο επικίνδυνη από την πολιτική συνιστόσα. Εμείς κάναμε και διάφορε ονοησίε ε, όταν έγινε η επίθεση στο Ιράκ ε, λόγω της ε, έλλειψης γνώσης του πολιτισμού έδωσε τη δυνατότητα σε μια σουνητική χώρα να ορίσει ΣΥΙΤΗ πρωθυπουργό ο οποίο έδωσε προνομία στη δική του κοινότητα μετά από την κατάρρευση του Ιρακινού στρατού από μισθοφόρους όπως έγινε σε όλες τις αραβικές χώρες για τους παλιούς δικτάτορες είχαμε το φαινόμενο μιας τεράστια ανεργία. Ανεργία που μεταφράστηκε στη συμμετοχή στον ΤΕΣ. Ε, και στον διάδοχο της Αλκάιντα. Πρόκειται για ανθρώπους ανέργους αλλά και χωρίς ελπίδα. Αυτή είναι η δική μου εξήγηση και αυτού του είδους την γενικευμένη ριζοσπαστικοποίηση ε, γενικευμένη ανησυχία την οποία παρατηρούμε σήμερα. Το θύμα της οποίας πληρώνουμε στην Ευρώπη. Γιατί όσοι διαπράξαν τις ε, επιθέσεις στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες ήταν άνθρωποι χωρίς ελπίδα που ριζοσπαστικοποιήθηκαν για κοινωνικούς λόγους. Η ριζοσπαστικοποίηση αυτή είναι ακόμα εντονότερη όταν ε, οι επικοινωνίες είναι πιο γρήγορες ε, Ε, θέλουμε κάποιες απαντήσεις για αυτά τα ζητήματα, αλλά ε, γυρίσουμε στο στρατιωτικό σκέλος ε, για τη σταθεροποίηση της περιοχής με την παρουσία του ΝΤΕΣ. Χρειάζεται μια πολιτική απόφαση για το Ιράκ. Τι γίνεται στο Ιράκ. στη Συρία η κατάσταση είναι να ενταθεί. Δεν έχουμε ένα πραγματικό κράτος στο Ιράκ θα λέγαμε ότι το κράτος έχει ε, πέσει, ε, υπάρχει πολυπολιτισμικότητα, εκατομμύρια άνθρωποι ε, που ανήκουν σε εθνικές ομάδε και υπάρχει μια άρνηση να εξευρεθεί λύση για τον πληθυσμό των Κουρδών. Κάτι που υπονομεύει την ασφάλεια στην περιοχή. αν βρούμε μια απάντηση για το Ιράκ, τότε θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε με τη Συρία. Θυμάμαι ότι εδώ στο Κοινοβούλιο, στην προηγούμενη θητεία, πόσοι Σύριοι πολεμιστές ε, έρχονταν στις Βρυξέλλες ζητώντα ε, υποστήριξη. Αλλά όλοι, σχεδόν όλοι, υποστήριξη θεωρούν τα όπλα, όχι την ε, διπλωματία, όχι την πολιτική. Όλοι ζητούσαν όπλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, η μόνη λύση πιστεύουμε θα είναι διπλωματική. Ε, όταν ε, ρίχνουμε βόμβες υπάρχει κίνδυνος να πλέξουμε τους πολίτες, τον άμαχο πληθυσμό και αυτό υπάρχει περίπτωση να οξύνεται η ροζοσπαστικοποίηση στην περιοχή. Συμφωνώ με τον καθηγητή κ. Βαλίεφ. Κατά την άποψή μου, ο Νότιος Κάφκασος, με εξαίρεση την Αρμενία, η οποία δεν έχει κανένα πρόβλημα ε, για, σε αυτόν τον τομέα. Η Γεωργία και το Αζερβαϊτζάν μπορούν να θεωρηθούν ε, περιοχές διέλευσης, αλλά είναι σταθερές, κοσμικές χώρες. Έχω μια ερώτηση λοιπόν προς εσάς. Αναφερθήκατε στη στάση της κυβέρνησης του Αζερμπαϊτζάν ε, ως προς τους ανθρώπους που επανέρχονται από τα πεδία μάχης της Συρίας, του Ιράκ άλλων περιοχών. Εσείς ε, έχετε ορίσει ως ποινικό αδίκημα τη συμμετοχή αζέρων ε, πολιτών σε τρομοκρατικές οργανώσεις ε, στις διαμάχες της Μέσης Ανατολής. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε. Γιατί όλοι συνηθίζουν να μιλάνε για ριζοσπαστικοποίηση, για πατριωτικές πράξεις, για πατριωτικό ζήλο, αλλά εγώ πιστεύω ότι μια ισχυρή αντίδραση στον τομέα του ποινικού δικαίου θα μπορούσε να αποτελέσει μια λύση και για τους Ευρωπαίους. Κατά την απόψή μου φυσικά. Ένα άλλο ερώτημα ε, προς την Φλωρόνς. Η κατάσταση της Συρίας υπάρχει κίνδυνος να εξαχθεί στη Λιβύη. Η Λιβύη είναι ένα ε, κράτος το οποίο έχει καταρρεύσει, δεν υπάρχει κυβέρνηση, παρότι αναφερόμαστε σε αυτήν ως κράτος. Υπάρχει περίπτωση να χρησιμοποιηθεί ως έδρα του όταν ε, η Διεθνή Συμμαχία τους ε, αναγκάσει να φύγουν από τη Συρία. Ποια είναι η απόψη σας γι' αυτό. Σε αυτό να προσθέσουμε τις ριζοσπαστικές δομές του Μαλή και του Νίγηρα και την αναφέρουμε στην Ποκοχαράμ εδώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Μπουστινάρου. Να σα ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε, είναι πάρα πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση. Το πρόβλημα όμως τι θα γίνει με το περιεχόμενο αυτής της συζήτησης εκτός της αιτούσης αυτής και πόσο θα μπορέσουμε να επηρεάσουμε την αποτελεσματικότητα των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξέροντας ότι δεν ανταποκρινόμαστε στις πραγματικές προκλήσεις που έχουμε ενώπιον μας. Πρώτο ερώτημα, μήπως πρέπει να αλλάξει την, τις πολιτικές που ακολουθεί η Ευρώπη για τις χώρες της Μεσογείου. Πόσο πρέπει να πώς πρέπει να κανονίσουμε το μείγμα αυτό της ασφάλειας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά. Η Ευρώπη είχε πάντα την τάση να φέρεται πατερναλιστικά προς τις χώρες αυτές και ένα δεύτερο ερώτημα, ξέρω ότι δεν είναι εύκολο αυτό το ερώτημα, αλλά είναι δύσκολη η καιρή και πρέπει να είμαστε λίγο πιο πραγματιστικοί. Αναφερθήκατε στη Λιβύη. Όλοι ξέρουν ότι η Λιβύη σήμερα γίνεται ένα καταφύγιο για πολλούς μαχητές. Μα είναι ήδη η Λιβύη μια χώρα διέλευσης για την περιοχή του Σαχέλ. Ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος λοιπόν μου έχουν πει πολλοί από το πολύ αξιωματούχοι και του Μαρόκου ότι είναι τόσο επισφαλής η σταθερότητα της περιοχής που μπορεί το Ισλαμικό κράτος να έχει πολύ έντονο αντίκτυπο στο Σαχέλ και το Νότιο Σαχέλ αν υπάρξει περαιτέρω αστάθεια. Δεύτερο ερώτημα, τι είδου συνεργασία θα πρέπει να κάνουμε με την Αίγυπτο, την Ιορδανία, το Μαρόκο και την Αλγερία, γνωρίζοντας ότι όλα αυτά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα ήταν ουσιαστικά μονοδρομικού χαρακτήρα. Αναφέρομαι σε κάτι που μου είπε ένας ηγέτης της περιοχής. Ακόμα και η παροχή, η συνεργασία μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών είναι μονόδομος από τις χώρες αυτές προς την Ευρώπη, αλλά όχι από την Ευρώπη προς τις χώρες αυτές. Η Ευρώπη κρατάει ένα εγωιστικό χαρακτήρα και δεν θέλουμε να μοιραζόμαστε τα στοιχεία που συλλέγουν οι δικέ μα υπηρεσίε πληροφοριών, ακόμα και μέσα στην ίδια την Ευρώπη. Λοιπόν, ποιο πρέπει να είναι ο ρόλο τη συνεργασία μα στα θέματα ασφάλειας με το Ισραήλ, που για να είμαστε ειλικρινεί έχουν πολύ μεγάλη συσσωρευμένη εμπειρία στα θέματα αυτά. <clears throat> Πιστεύω ότι η εμπειρογνωμοσύνη που έχει συλλέξει το Ισραήλ θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σημαντικές για να μας βοηθήσει να φτιάξουμε ένα μοντέλο αντιμετώπισης, όχι ακολουθώντας το παράδειγμα του Ισραήλ κατά ανάγκη, αλλά να βρούμε έναν τρόπο στο ευρωπαϊκό έδαφος να μην έχουμε να κάνουμε με μεγάλης κλίμακος τρομοκρατικής, τρομοκρατικές επιθέσεις, γιατί ήδη καταμετρούμε νεκρούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε ανησυχητικό επίπεδο. Και τέλος, επειδή ορθά αναφερθήκατε στο θέμα της αντιμετώπισης των χωρών αυτών, πώς θα τις ανοικοδομήσουμε μετά τον πόλεμο. Δεν έχουμε στρατηγική ούτε για την Συρία, ούτε για το Ιράκ. Αυτό είναι απαράδεκτο και ασυγχώρητο, γνώριζοντας ότι οι άνεργες στρατιωτικές ελίτ θα κάνουν αυτό το οποίο ξέρουν καλύτερα να κάνουν. Θα πολεμήσουν και πάλι, θα φτιάξουν συμμορίες, ομάδες, θα μπουν σε παράνομες και εγκληματικές ενέργειες. Εμείς ανοήτως δεν το λάβαμε αυτό υπόψη στο Ιράκ. Λοιπόν, αυτό το οποίο πρέπει να κάνει, τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει η Ευρώπη για να αντιμετωπίσει τις χώρες αυτές μετά από την κατάπαυση του πυρός, μετά από την πάυση των εχθροπραξιών, να δώσει δυνατότητες ανάπτυξης, να αλλάξει το επικρατούν. Παράδειγμα, ώστε οι πληθυσμοί να θέλουν να παραμείνουν εκεί. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις. Και θα ήθελα επίσης να αναφερθώ και στους πολέμους δι αντιπροσώπων. Αυτές οι συγκρούσεις ουσιαστικά έχουν υποστηριχθεί από ορισμένου μέσα σε εισαγωγικά επενδυτέ, οι οποίοι τυχαίνει να είναι κάποιοι από αυτούς και εταίροι της Δύση. Εμεί θεωρούμε ότι αυτό δεν είναι πρόβλημα δικό μου, αν μπορώ να πουλήσω περισσότερα όπλα στους εταίρους μου, αυτό είναι καλό. Καλή δουλειά είναι αυτή. Αλλά φυσικά όλα αυτά στρέφονται ως μπούμερανγκ εναντίον μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν για, την, ε, για τις ε, ανακοινώσεις σας και θα ήθελα να έχω και την εγγραφή μορφή των ε, παρεμβάσεων σας ή δυνατόν να απαντήσω σε αυτό που είπατε κύριε Μποστινάρου Να Βέβαια δεν, είναι, δεν νομοθετεί η Επιτροπή μας, κυρίως ε, οι συζητήσεις που έχουν ενδιαφέρον με ειδικού που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, αυτό είναι το βασικό μας εργαλείο. Α, θα δείτε ότι εδώ έχουμε πληθώρα επισκεπτών, παρατηρητών που μας παρακολουθούν Επίσης ε, προβάλλεται και στο διαδίκτυο η συζήτηση και ξέρω ότι μας παρακολουθούν ε, πολλοί. Ε, αυτό είναι καλό. Έχουμε κάποια επιρροή δηλαδή στην εξέλιξη των πραγμάτων. Με αυτή την ευκαιρία ήθελα να κάνω δύο σκέ... μερικές σκέψεις και να κάνω ερωτήσεις και στους δύο μιλητές. Ε, να ευχαριστήσω την κυρία Φλωράνς Γκάουμπ καταρχήν για την εξαιρετική παρουσίαση. Συμφωνώ με τον ε, κύριο Φρόιν που θυμήθηκε την πρώτη φορά που βρεθήκαμε. Σίγουρα η Λιβύη είναι κάτι παραπάνω από ορατή ως πιθανός τελικός προορισμός των μαχητών του Άισις λόγω κάποιων χαρακτηριστικών ουδετερότητας αυτής της χώρας που είναι τόσο κατακαιρματισμένη. Ε, υπάρχουν υπάρχουν πολλές κοινότητες, ε, πολλά κομμάτια του πληθυσμού, ομάδες ε, που θέλουν να αναζωπηρώσουν το παρελθόν τους. Θέλω λίγο να αντιστρέψω την ερώτηση του κυρίου Φρόιντ. Κατά πάσα πιθανότητα, και από ό,τι παρατηρώ, ε, αυτή, αυτές οι διάφορες ε, ε, εθνοφυλακές που αναπτύσσουν δράση δρούν ε, ανασχετικά σε σχέση με την επιτυχή κατάληξη μιας πολιτικής διαδικασίας. Είναι μια μορφή έμεση διείσδυση. Τι χρονικά περιθώρια έχουμε για να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία και πώς θα περιγράφατε τη δυναμική της. Υπάρχουν κάποια γρήγορα ωφέλη, όπως γνωρίζουμε, σε σχέση με κάποιες πρόσθετες δυνατότητες χρηματοδότησης της ΆΙΣΙ στην ε, Λιβύη. Πώς έχει το θέμα εκεί. Ερώτηση και προς τους δύο ομιλητές. Πώς έχει η κατάσταση μεταξύ των, της Ιητικής και Σουνητικής κοινότητας και τι εντάσεις υπάρχουν σε διάφορες περιοχές, γιατί ξέρω ότι και αυτή είναι σημαντική συνιστόσα που επηρεάζει την όλη κατάσταση. Ίσως ε, ε, είναι, ε, δεν είναι τόσο επικίνδυνο όσο στο Αζερβαϊτζάν αλλά στη Γεωργία υπάρχουν ήδη εντάσεις. Και ε, η κοινότητα που απειλείται περισσότερο είναι η κοινότητα των χριστιανών, γιατί υπήρξαν αρκετά περιστατικά πραγματικών απειλών ε, εναντίον της κοινότητας αυτής. Λοιπόν, οι ομιλητές μας θα απαντήσουν. Ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά τα σχόλια και τις ερωτήσεις. Ε, ακολουθώ τις σημειώσεις μου. Ε, πριν από 1,5 χρόνο για το Ιράκ φαντάζομαι ότι θα είχα πει τα ίδια πράγματα, διότι δεν έχουν ε, αλλάξει πολλά από τότε σε αυτό το μέτωπο. Ε, αναφέρατε κάτι πολύ ενδιαφέρον, η ψυχολογία του ISIS, η ψυχολογία βίαιων ομάδων, δηλαδή πώς λειτουργούν στη στρατολόγηση και ε, διατήρηση των μελών τους. Αυτό που είναι ενδιαφέρον στο ISIS είναι ότι είναι ένα μείγμα, ε, έλαβε οικονομικά μαθήματα από εγκληματικά δίκτυα, δηλαδή όταν πρόκειται για εκβιασμούς, απαγωγές κλπ. Αλλά όταν πρόκειται για διαχείριση προσωπικού, ε, έμαθε πολλά από εκεί. Υπάρχει λοιπόν μια ψυχολογική διάσταση που έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή διάσταση του ISIS. Όταν είναι νέος, ε, Ιρακινός, Ισύρος κλπ. Μπορεί να ε, έχει διαφορετικά κίνητρα. Αλλά υπάρχουν και τα ευρωπαϊκά κίνητρα, τα κίνητρα των Ευρωπαίων. είδαμε ότι οι τρομοκρατικές ε, ομάδες ε, ε, έχουν παρόμοιους τρόπους στρατολόγησης. Τα κοινωνικά μέσα έχουν ταχύνει αυτή την κατάσταση. Δηλαδή αυτός που στρατολογεί εντοπίζει έναν άνθρωπο που έχει κάποιες συμπάθειες, αλλά μετά παρακολουθεί το ψυχολογικό του προφίλ, βλέπει τα κίνητρα, τα οποία μπορεί να είναι τέσσερα, μπορεί να είναι τυχοδιοκτισμός, μπορεί να είναι ανθρωπιστικά κίνητρα, μπορεί να είναι διάφορα. Μετά τι γίνεται. Αυτό δεν αρκεί. Θα πρέπει να υπάρχει μια αίσθηση απώλειας στη ζωή ενός ανθρώπου για να είναι δεκτικό σε τέτοια μηνύματα. Και αυτή η απώλεια μπορεί να πάρει διάφορες μορφές. Μπορεί να είναι απώλεια σχέσης, απώλεια γονιού, απώλεια θέση εργασίας, απώλεια κατοικίας. Κάτι λείπει από τη ζωή του ανθρώπου. Και μετά η θρησκευτική έρωση, η τρομοκρατική οργάνωση μπαίνει και γεμίζει το κενό με νόημα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Βέβαια, μια επιτυχής οργάνωση, όπως είπατε, ε, εξελίσσεται εκθετικά. Γιατί συνήθως μπαίνει κανείς σε μια οργάνωση που είναι ήδη μεγάλη και αυτό επικυρώνει την επιλογή, την ε, ατομική επιλογή. Νιώθει κανείς καλύτερα όταν μπει σε μια μεγάλη οργάνωση που έχουν μπει πριν από σένα κι άλλοι πολλοί από την άλλη όταν χάνει μια οργάνωση στο πεδίο μάχης, χάνει ως ένα βαθμό και μέλη. Αλλά η ψυχολογική βοήθεια, η αίσθηση του ανήκειν, της κοινότητας των φίλων αυτό εξακολουθεί να υφίσταται. Αυτοί, κάποιοι που έχουν φύγει από κάποια αίρεση εξακολουθούν να είναι ε, δεκτικοί. Δηλαδή σε λανθάνουσα κατάσταση ανταποκρίνονται. Δεν ισχύει αυτό στον ίδιο βαθμό για όλους, αλλά ο πρώτος κανόνας είναι ότι αν έχει ε, μπει κανείς, αν έχει υπάρξει μέλος για πάνω από ένα χρόνο σε θρησκευτική ή τρομοκρατική οργάνωση, είναι δύσκολο να αναστραφεί αυτή η ψυχολογική αίσθηση του ανήκειν. Καταστροφή του ISIS λοιπόν δεν θα σπάσει κατά ανάγκη τους δεσμούς των μελών που έχουν διαμορφωθεί. Δεν λέω ότι θα γίνουν όλοι τρομοκράτες, αλλά υπάρχει ένα δίκτυο το οποίο γεννήθηκε ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Το άλλο πιο ανησυχητικό είναι ότι για να ε, ε, γίνει ένα τρομοκρατικό πλήγμα όπως στις Βρυξέλλες στο Παρίσι. Αυτό είναι πολύ φθηνό. Δεν χρειάζονται πολλοί άνθρωποι, ούτε χρειάζονται πολλά χρήματα για να γίνει μια τέτοια επίθεση. Με 10.000 ευρώ μπορεί να καλυφθούν ε, έξοδα μεταφοράς, το υλικό αυτά αγοράζονται και από ένα φαρμακείο ή σε ένα σούπερ μάρκετ. Ε, ε, ε, δεν χρειάζονται για ένα πλήγμα από πολλά δύσκολα πράγματα. Και αυτό είναι σημαντικό. Κάτι άλλο είναι ότι ακόμα και αν πεθάνει το ISIS, η μέθοδος και η ιδέα θα επιβιώσει αν δεν αντικατασταθεί από άλλα μέτρα. Πριν από την ISIS είχαμε την Αλκάιντα και η Αλκάιντα εξακολουθεί να είναι ενσωή. Δεν την πολύ συζητάμε τώρα, αλλά είναι πολύ δραστήρια. Δεν έχει εξαφανιστεί ακόμη. Και ε, εγώ ανησυχώ διότι η εστίαση στο στρατιωτική συνιστόσα χρήσιμη μεν, αλλά όχι ικανή. Για τη Λιβύη Όλη η διαδικασία υπάρχει γιατί αναδύεται ένα θέμα ασφαλείας, αλλά ε, αυτές οι εθνοφυλακές στη Λιβύη ε, είναι πολύ ενδιαφέρουσες, γιατί δεν είναι συνεκτικές, ούτε μιλούν με μια φωνή όλες. Ε, πολλαπλασιάστηκαν μετά τη σύγκρουση, τουλάχιστον διπλασιάστηκαν, αν δεν είναι και παραπάνω, και δεν έχουν μια συνεκ, ένα ε, συνεκτικό θεματολόγιο, δηλαδή δεν δρούν είναι δραστήρια ε, συνολικά στις διαπραγματεύσεις. Αυτοί που διαπραγματεύονται δεν τους ελέγχουν, έχουν χαλαρές διασυνδέσεις, ε, αλλά ο καθένας εξυπηρετεί τα δικά του συμφέροντα και μετά το 2011, γι' αυτό ήταν πρόκληση η Λιβύη, γιατί είχαμε δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, αλλά η κυβέρνηση αυτή δεν ήταν απλούστατα ικανή να ασκήσει ε, πυροή και έλεγχο ε, σε όλους αυτούς. Ο Πρωθυπουργό πολλές φορές έλεγε ότι πάμε για αφοπλισμό τώρα, αλλά δεν γινόταν αφοπλισμός, γιατί κανείς δεν παρέδιδε τα όπλα. Είναι φαύλος κύκλος. Και αυτό δεν γίνεται μόνο στη Λιβύη, θεωρώ εγώ. Μετά από εμφύλιο, ο αφοπλισμός όλων αυτών θα πρέπει να στηρίζεται στην κοινωνική συνένεση και στη Λιβύη. Δεν έχουμε στρατιωτική οργάνωση ή δύναμη αστυνομική που θα μπορούσε να την κάνει αυτή τη δουλειά. Ε, βέβαια, ε, ο ισχυρισμό είναι ότι υπάρχει ο στρατό στη Λιβύη, αλλά έχει αποδεκατιστεί. Ε, και ο διοικητής ε, του τον Μπρούκ ε, παίζει ρόλο ε, κακό και ε, ανέφερε ότι ε, δεν εμπιστεύεται στους πολιτικούς που θα απασπρώξουν τη Λιβύη στην Άβυσσο και ε, την απειλή ε, ένοπλης βίας. Άρα λοιπόν ε, ο δεν ελέγχεται από το τον και έχει τη δική του πολιτική ατζέντα, άρα μπορεί να ε, καταρρύψει όλη τη διαδικασία να αποφασίσει. Ε, γι' αυτό είπα ότι όσοι ασχολούνται με την, το θέμα της ασφάλειας δεν καλύπτουν αυτή τη διαδικασία. Και ε, αυτό έχει να κάνει με την, ε, τον κατακαιρματισμό στα θέματα ασφαλείας στην Λιβύη. Να απαντήσω στα γαλλικά στην κυρία Νικολάη. Λοιπόν, είπατε ε, αυτή την πολύ ωραία ιδέα των τεσσάρων εποχών του Βιβάλντι. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι αυτά που βλέπουμε σήμερα στην περιοχή είναι μία μακροχρόνια ε, διαδικασία μετασχηματισμού. Δεν είναι δηλαδή μόνο φθινόπωρο ή χειμώνα. Παρατηρούνται πολλέ εποχέ πολιτικών μετασχηματισμών. Και παρότι αυτή τη στιγμή προκαλεί τεράστια δυστυχία, ε, είναι κάπω μοιραίο. Ε, έχουμε να αποκομίσουμε κάποια διδάγματα για την περιοχή από όλα αυτά πώς θα τους μιλήσουμε πολιτικά, ποιο είναι ο ρόλο των πολιτών, ο ρόλο του κράτου κτλ. Αλλά μία πτυχή που αναφέρατε στην οποία θέλω να εστιαστώ είναι ο πολιτικός αποκλεισμός. Αναφέρατε το Ιράκ, αλλά να σας δώσω τα νούμερα για να σας εξηγήσω πόσο δραματική είναι η κατάσταση στην περιοχή. Το ιστορικό παράδειγμα φυσικά είναι η Γερμανία μετά το 1945. Κοίταγα τα νούμερα. Πράγματι στη Γερμανία το 1% του πληθυσμού αποτέλεσε το αντικείμενο πολιτικών μέτρων αποκλεισμού. Η πρώην Αν σκεφτούμε ότι εκείνη την εποχή στη Γερμανία μια μικρή οικογένεια είχε δύο παιδιά ε, και δύο γονείς ε, και ένα οικονομικό περιβάλλον που επέτρεπε την εργασία και στον ιδιωτικό τομέα πρέα του δημοσίου. Στο Ιράκ τώρα συγκριτικά μετά το 2003 το 3% του πληθυσμού ε, υπέστη αποκλεισμό. Σκεφτείτε ότι συνήθω οι οικογένειε είναι μεγαλύτερε, έχουν τέσσερα παιδιά, έχουν συνήθω την ευθύνη και των ε, παππούδων, διότι δεν υπάρχει κοινωνικό σύστημα και το οικονομικό περιβάλλον δεν ε, δίνει και δυνατότητε εργασία στον ιδιωτικό τομέα. Αλλού οι περισσότερε θέσει εργασία στην ειρηνική οικονομία είναι στο δημόσιο. Οπότε μιλάμε για το άνω του 10% των ατόμων αν χάσει κάποιο τη δουλειά του, δεν μπορεί να πάει να δουλέψει αλλού. Στη Λιβύη, ε, το ξεχνάμε συχνά, ο νόμος πολιτικής απομόνωσης ψηφίστηκε το 2013 και βλέπει πολλά περισσότερα από ότι παρόμοιοι νόμοι αλλού αφορά το 10% του πληθυσμού της Λιβύης ε, και σκεφτείτε πάλι πόσο μεγαλύτερες είναι οι οικογένειες Στη Λιβύη, ξέρετε, η οικονομία είναι ακόμα λιγότερο ε, ε πολυπίκυλη από ό,τι στο Ιράκ. Ε, η συντριπτική πλειοψηφία των θέσεων εργασία είναι στο δημόσιο. Αν δεν εργαστικά στο δημόσιο, δεν έχει να πάει πουθενά άλλο. Και αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, ειδικότερα στο Τουμπρούκ, όπου άνθρωποι υφίστανται αποκλεισμό χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τι έκαναν το 2011, αν άλλαξαν άποψη και τι έκαναν πριν. Αποκλείομαστε, δηλαδή, αποκλείεται δηλαδή κανείς αυτόματα αν έχει εργαστεί στο προηγούμενο, υπό το προηγούμενο καθεστώς. Ακόμη και αν ήταν βιβλιοθηκάριος ε, ή εργαζόταν σε ένα ερευνητικό ίδρυμα. Απομονώνεται από το σύστημα χωρίς ε, δεύτερο λόγο και αυτό παίζει σημαντικό ρόλο, ενώ συχνά το ξεχνάμε. Και κάτι τελευταίο, αναφέρατε τη Συρία, οι λύσεις ε, για τη Συρία βρίσκονται εντός της Συρίας οι αεροπορικές επιδρομές δεν πρόκειται να επιλύσουν το πρόβλημα πιθανότατα. Χρειάζεται μια ε, συριακή πολιτική λύση που θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα πριν το 2011. Δηλαδή το πρόβλημα σήμερα δεν είναι ο ΣΑΝΤ ή το ISIS, είναι η δυσαρέσκεια εντός του ε, πληθυσμού της Συρίας, ήδη με το προηγούμενο καθεστώς. Και τέλος, τι θα κάνουμε τώρα. Ε, αναφέρετε τα πιο ακαθόδη ζητήματα σε ερωτήσεις και είμαι εδώ για να σας βοηθήσω να βρείτε κάποιε απαντήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι καλό ε, στο να ενισχύει την ευαισθητοποίηση. Ε, μπορεί να πει πράγματα που άλλοι υπεύθυνοι χαρακτηριστικοί πολιτική δεν δίνονται να πούν. Νομίζω το πρώτο είναι ότι πρέπει να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε ότι έχουμε επιλογή μεταξύ ασφαλεία και ανθρώπινων δικαιωμάτων. Μπορεί να υπάρχει συνεργασία, ανταλλαγή ε, πληροφοριών και ταυτόχρονα να παρέχονται και ανθρώπινα δικαιώματα επαρκεί. Επίσης τα πράγματα δεν είναι απλά. Οι χώρες με κακό ιστορικό ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι οι πιο ε, επικίνδυνες. Η Αλγερία που έχει να προσφέρει πολλά. Η, η Αλγερία ε, έχει πολλά να προσφέρει και δεν θέλουμε να ακολουθήσει την οδό των άλλων χωρών. Οπότε εμεί υποστηρίζουμε μεγαλύτερη συνεργασία με την Αλγερία. Οπότε εδώ, ειδικότερα στο Κοινοβούλιο, δεν πρέπει να ε, ακολουθείτε αυτή την οδό τη κατορμασία ορισμένων χωρών. Αυτό που ε, αξίζει, το είπε η κυρία Νικολά, έχουμε το χώρο Σέγγεν. Και έχουμε και το παράνομο Σέγγεν, όπως λέγεται. Δηλαδή, Ε, ξέρετε, άτυπα μπορεί να περάσει κανείς τα σύνορα από το Μαρόκο στην ε, Αλγερία και μετά να περάσουν στη Λιβύη και έχει πολλούς Μαροκινούς ε, μαχητές που έχουν περάσει στη Λιβύη. Είναι μια δύσκολη περιοχή προς παρακολουθήσεις για γεωγραφικούς λόγους. Η Αλγερία έχει κλείσει μεν όλα τα σύνορα, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, προσπαθεί να σταματήσει να εμποδίσει και την Τινησία να πέσει στην ίδια παγίδα, αλλά ισορροπία, αν θέλουμε μακροχρόνια σταθερότητα, ε, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με αντιμετώπιση και των δύο πτυχών της ασφάλειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή, μάλλον ε, θα έλεγα τα θεμελιώδη πράγματα που πρέπει να προσφέρει ένα κράτος, την ευημερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, το, ε, την ευημερία, όλα αυτά. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο στη στρατηγική για μετά τη διένεξη. Δεν είχαμε τέτοια στρατηγική στο Ιράκ και στη Λιβύη, αλλά κάτι σημαντικό πιστεύω, κάτι που, στο οποίο μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς ως ε, εκπρόσωποι των πολιτών, είναι να ενημερώσετε το κοινό ότι οι στρατηγικές ε, για τις ε, περίοδους μετά τις διενέξεις χρειάζονται πολύ χρόνο, τουλάχιστον μια δεκαετία, χρειάζονται χρήμα, αλλά στο απότερο μέλλον αποδεικνύονται φθηνότερες ως λύσεις. Εμεί προσπαθούμε τώρα να κάνουμε μια τέτοια μελέτη με διάφορα υποθετικά σενάρια. Τι θα είχε γίνει αν είχαμε φτιάξει τα πράγματα στη Λιβύη αμέσω μετά από την πάυση τη διένεξη. Θα ήταν κάτι που δεν θα ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή σήμερα, αλλά δεν θα είχε οδηγήσει τα προβλήματα, θα είχαμε αποφύγει τα σημερινά προβλήματα. Γιατί ξέρετε, ο κόσμο σήμερα θέλει να επιλέγει τα προβλήματα σε έξι μήνε, αλλά αυτό δεν γίνεται τόσο εύκολα. Σε ολόκληρη την περιοχή πριν περάσω στους Σουνιτές και τους Σιήτες, που είναι το τελευταίο μου σημείο, χρειαζόμαστε οικονομικό εξυγχρονισμό. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε συνεργαστεί πολύ με όλες τις χώρες της περιοχής. Ε, σημαίνει τεράστια ανάπτυξη το εμπόριο μεταξύ Ευρώπης. Αυτό είναι καλό. Αλλά οι δομές τους δεν είναι εξυγχρονισμένες ε, όσον αφορά τη γεωργία, για παράδειγμα. Έχουν το προσωπικό που θέλουν, έχουν τους νέους ανθρώπους που χρειάζεται για τον εξυγχρονισμό αλλά υπάρχουν αυτές οι αποπνικτικές παλιές δομές που δεν λειτουργούν. Έχουμε μια έκθεση της Παγκοσμίας Τράπεζας για την Τινησία που δείχνει ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια απελευθέρωση των ε, δικτύων και της τηλεφωνίας, ε, των αερομεταφορών, ε, πράγματα που δεν συνέβησαν για πολιτικούς λόγους. Κάτι τελευταίο για τους και τους Σιήτες. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα τεράστιο αλλά νέο υπό τη σημερινή του μορφή. Πριν 20 χρόνια δεν είχε τη μορφή που έχει σήμερα, οπότε αυτό δεν κακό. Είναι καλό ότι ε, να ξέρουμε ότι δεν θα έχει την ίδια μορφή επάπειρων, αλλά έχουμε ε, την προσέξη από ε, μεταξύ φατριών από πάνω προς τα κάτω έχουμε τη Σαουδική το Ιράν από τη μία και από την άλλη το Χεσμπολά όλους αυτούς που παίζουν αυτό το χαρτί της ε, φατρίας Αυτά, ξέρετε, ευδοκιμούν σε μέρη όπου ο κόσμος αισθάνεται ότι το κράτος δεν τον υποστηρίζει. Ε, και έτσι χρειάζεται να πάει να ψάξει αλλού θέσει εργασία και ασφάλεια. Οπότε, τίθεται πάλι ζήτημα αντοχής και σταθερότητας του κράτους. Το κράτος που πρέπει να παρέχει. Ε, στη στρατηγική λοιπόν θα εξετάσουμε αυτή την αντοχή του κράτους για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα. Και πάλι αυτό απαιτεί πολύ χρόνο. Δεν απαιτεί μόνο συνεργασία σε θέματα ασφαλεία. αλλά τίθεται ξανά το ζήτημα αυτό. Ποια είναι η φύση ενό κράτου ποια είναι η δουλειά του κράτου. Το κράτο λοιπόν η δουλειά του είναι να παρέχει ευημερία, εκπροσώπηση, ενδεχομένω, ασφάλεια και να αποτελεί δημοσιολαβητή μεταξύ των διαφορών ομάδων που ζουν εντό του κράτου αυτού. Και όταν το κράτο υπολείπεται των υποχρεώσεών του, τότε ε, οδηγούμαστε στις ε, άλλε καταστάσει φυσικά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της ε, ποινικοποίηση των ε, ανθρώπων που βρέθηκαν σε χώρες όπου πολεμήσαν ως ξένοι μαχητές. Υπάρχει μεγάλη, μεγάλο ιστορικό στο Αζερμπάτζαν και στη Γεωργία για τους μαχητές αυτούς είναι ο ίδιος φόβος που είχε η Σαουδική Αραβία το 1980 όταν πήγαν Μουτζαχεντίνα από τη Σαουδική Αραβία στο Αφγανιστάν, πολέμησαν, νίξαν τους Ρώσους και μετά γύρισαν στις χώρες τους. Και έτσι ουσιαστικά ξεκίνησε όλη η ιστορία της Αλκάιντα λόγω του πολέμου κατά το, της Σοβιετικής Ένωσης. Είναι κάτι που απασχολεί ιδιαίτερα τις χώρες αυτές όπως η Γεωργία και η Αζερμπαϊτζάν. Ξεκινώντας από την δεκαετία του 1990 όταν πήγαν οι πρώτοι μαχητές στην Τσετσενία και πολέμησαν κατά τον Ρώσο, αυτή ήταν η πρώτη εμπειρία που είχαν και οι δύο κυβερνήσεις όταν έχασαν τον, τον πόλεμο με τους Ρώσους στην Τσετσενία, οι πιο πολλοί από αυτούς γύρισαν στις πατρίδες τους και επομένω σε αυτή την κατάσταση υπήρξε ο κίνδυνο ότι θα χρησιμοποιούσαν τις δεξιότητες αυτοί οι άνθρωποι και τις διασυνδέσει του για να δημιουργήσουν διαταραχές στην κυβέρνηση. Η, κυβέρνηση του Αζερβαϊτζάν πήρε κάποια δρακόντια μέτρα για να σταματήσει αυτή την πιθανότητα και υπήρξε πομπινικοποίηση και βαριέ ποινέ για αυτού οι οποίοι είχαν πάει κάπου αλλού. Ένας, ε, ένα άτομο που κατηγορείται για τρομοκρατία μπορεί να πάρει 8 ή 9 χρόνια φυλακή, αλλά ένας ε, που έχει υπάρξει ξένος μαχητής κινδυνεύει με 14-16 χρόνια. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος ότι αυτοί που ήταν σε μια τρομοκρατική οργάνωση στο παρελθόν μπορούν να θεωρηθούν ότι προσπάθησαν να ανατρέψουν την κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν. Είναι αλήθεια ή όχι, δεν το ξέρουμε, αλλά γι' αυτό είναι αυξημένες οι ποινές που επισύρει αυτή η ιδιότητα του ξένου μαχητή. Θα προτιμούσα λοιπόν να τους θεωρήσουν μονάχα τρομοκράτες παρά ξένους μαχητές. Αυτό ήταν ο λόγος λοιπόν για την ποινικοποίηση των ενεργειών αυτών των μαχητών. Και επομένως υπήρξαν κάποιες μικρές ομάδες οι οποίες γύρισαν από τη Συρία και το Ιράκ και υπέστησαν αυτές τις βαριές κυρώσεις. αλλά εδώ υπάρχει και μια κάποια παρανόηση του ρόλου του Ισλαμικού κράτους. Πολλές κυβερνήσεις και όχι μόνο το Αζερβαϊτζάν παρεξηγούν το γεγονός ότι το Ισλαμικό κράτος δεν είναι ο διάδοχος της Αλκάιδα. Είναι ένα τελείως διαφορετικό είδος οργάνωσης, ούτε καν οργάνωσης δεν θέλω να πω, γιατί δεν έχει τον ε, κλασικό χαρακτήρα μια οργάνωσης που έχει ένα ηγέτη, ενεργού υποστηρικτέ και παθητικού υποστηρικτέ. Δεν έχει αυτή τη μορφή οργάνωσης. Και επίση η Αλκάιδα ποτέ δεν θέλησε να πει ότι εμείς θέλουμε να έχουμε ένα δικό μας έδαφος. Ήταν μια τυπική αστικού πολέμου οργάνωση η οποία ήθελε να κάνει καταστροφές, τρομοκρατικές ενέργειες και μετά να αποσυρθεί χρειάζεται για να το κάνει αυτό να έχει πολλά θύματα και όλα αυτά, αλλά ποτέ δεν θεώρησε ότι ήθελε να έχει μια εδαφική βάση, ενώ το Ισλαμικό κράτο προσπαθεί να καταλάβει έδαφο και να έχει μια επικράτεια που να την ελέγχει. Ξεπερνάει λοιπόν την Αλκάιδα, έχει ένα έδαφος το οποίο είναι το χαλιφάτο του, έχει μια παρουσία στο διαδίκτυο. Όλα αυτά η Αλκάιντα δεν τα είχε και γι' αυτό δεν είχε τόσους πολλούς που να τους προσιλητήσει. Είναι πάρα πολύ πιο ελκυστικό λοιπόν το σύστημα του Ισλαμικού Χαλιφάτου ή του Ισλαμικού κράτους για όλα αυτά τα άτομα τα οποία, σύμφωνα με τους συναδέλφους μου, είναι απόκληροι οικονομικά ή κοινωνικά ή πολιτικά ή αυτούς που περνάνε από μια κρίση ταυτότητας για πολλούς από τη Γεωργία και το Αζερβαϊτζάν που πηγαίνουν στο Ισλαμικό κράτος και σε άλλες αλαφιστικές ομάδες είναι τα άτομα που έχουν περάσει στο παρελθόν μια κρίση ταυτότητας. Γιατί έχουν αυτή την κρίση ταυτότητας. Γιατί πρώτα απ' όλα μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης δεν είχε αναδειθεί καμία νέα ιδεολογία στην περιοχή αυτή. <clears throat> Πηγαίνετε στο Νότιο Κάφκασο, στη Ρωσία, στις Σοβιετικές χώρες, στα Βαλτικά κράτη. Βλέπετε ότι υπάρχει ένα κενό ιδεολογίας δεν υπήρξαν δημοκρατικές ιδέες οι οποίες να ριζώσουν ο εθνικισμός κάπου βρέθηκε στο περιθώριο και επομένως η θρησκεία ως στοιχείο ταυτότητας, στη θρησκεία ως πηγή ριζοσπαστικοποίησης είναι μια πολύ ελκυστική ιδέα βγείτε από αυτό το χώρο, ελάτε στο δικό μας έδαφος του Ισλαμικού κράτους και θα σας δώσουμε μια νέα ζωή. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλούς οι οποίοι πηγαίνουν στο έδαφος του Ισλαμικού κράτους με τις οικογένειές τους, με τα μικρά τους παιδιά και μένουν εκεί. Δεν είναι όλοι μαχητές, θέλουν να ζήσουν όμως στο χώρο του Ισλαμικού Καλυφάτου. Και αυξάνεται ο αριθμό αυτών των ανθρώπων, όχι μόνο στο Αζερβαϊτζάν και στην Γεωργία, αλλά και στην Ευρώπη. Πολλοί από αυτού που πήγαν εκεί δεν πήγαν για να πολεμήσουν. Πήγαν για να ζήσουν σε ένα χώρο που καλύπτει την κρίση ταυτότητά του. Είναι δεύτερη γενιά μετανάστε, δεν έχουν καμιά σχέση με την τοπική κοινωνία. Και αυτό είναι ένα πραγματικό θέμα για μια πιο λεπτομεριακή κοινωνιολογική συζήτηση. Για την διαμάχη των Σιητών με τους Σουνίτες στην περιοχή του Νότιου Καυκάσου δεν υπήρξε ποτέ, δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα όπως υπήρξε στο Πακιστάν, στο Ιράκ, στη Συρία γιατί η κυβέρνηση είχε μεγάλη εξουσία και αυστηρό έλεγχο που δεν επέτρεπε να υπάρχει λειτουργία εσωτερικών οργανισμών, οργανώσεων που βασιζόντουσαν στη θρησκεία. Δεν τους άφησε να λειτουργήσουν εκεί. Αλλά, όσο και να μην το θέλουμε, πρέπει να επενέσουμε λιγάκι και τις Ιρανικές αρχές, οι οποίες δεν όθησαν σε κλιμάκωστη κατάσταση στη Γεωργία ή στο Αζερβαϊτζάν, δεν ποτέ δεν θέλησαν να ξεσπάσουν την οργή τους σε βάρος του πληθυσμού των ε, Σουνιτών. Δεν ενδιαφέρεται το Ιράν λοιπόν στο να αναμοχλεύσει σε βία στον Νότιο Καυκάσο. Και οι σαλαφιστικές οργανώσεις που είναι ενεργές στην περιοχή αυτή, οι πιο ριζοσπαστικές από αυτές μπορούν να είναι επικίνδυνες γιατί θα ανατρέψουν αυτή την ισορροπία μεταξύ των ομολογιών του Ισλάμ. Το Ισλαμικό κράτος λοιπόν στη Συρία, στο Ιράν, στο, στο Ιράκ, στο Νότιο Κάφκασο δεν θεωρεί ότι ο αντίπαλος του είναι οι χριστιανικές ή ιουδαϊκές <clears throat> κοινότητες, αλλά η κοσμική εξουσία και οι μουσουλμάνοι που δεν ακολουθούν τις δικές τους επιταγές, δηλαδή οι ΣΥΙΤΕΣ. Αυτοί φοβούνται λοιπόν θα είναι το, ο επόμενος στόχος του Ισλαμικού κράτους και όχι μονάχα τα κοσμικά καθεστώτα οι χριστιανικές και οι ιουδαϊκές κοινότητες των περιοχών. Οι χριστιανικέ και οι ιουδαϊκές κοινότητε λοιπόν στο Νότιο Κάφκασο δεν κινδυνεύουν τόσο πολύ όσο η κυβέρνηση και οι σιητικές κοινότητες εκεί. Ευχαριστώ πολύ λέγει η Πρόεδρος. Θα σα ζητήσω συγγνώμη γιατί κάπω ο κύριο Καστάλντο δεν μπόρεσε να λάβει το λόγο προηγουμένω, οπότε θα του δώσουμε σε ένα δεύτερο γύρο την δυνατότητα να λάβει το λόγο. Κύριε Καστάλντο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ζητήσω κι εγώ συγγνώμη στους προσκεκλημένους μας για την καθυστερημένη μου άφηξη και για τις ερωτήσεις μου ε, τόσο αργά. Θα συνεχίσω στα γαλλικά. Ευχαριστώ για την ευκαιρία και ζητώ πάλι συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ήθελα να κάνω κάποιες ερωτησούλες. Συμφωνώ με τα όσα είπε η κυρία Γκάουμπ για τον πολιτικό αποκλεισμό. Ορισμένες φορές δεν δίνουμε αρκετή σημασία σε αυτή τη συνιστόσα, ωστόσο υπάρχουν διαφορές μεταξύ Λιβύης και Ιράκ. Και στις δύο περιπτώσεις δεν θα μπορούσε το Ντάις να είχε κατασταθεί στην περιοχή αν δεν είχαμε αποκλείσει ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού από τη διαδικασία ένταξης στο Ιράκ. Μιλάμε για τη σουνητική κοινότητα και σκέφτομαι, το, έχω στο τώρα τον πρώην στρατό του Σαντάμα, ε, πως τόσο έδωσε τις γνώσεις και την εμπειρογνωμοσύνη στον ΤΑΕΣ για να χρησιμοποιεί συγκεκριμένα ιδιοπλισμού τα οποία διαφορετικά, στα οποία διαφορετικά δεν θα μπορούσε να είχε εκπαιδευτεί και όσον αφορά τη Λιβύη σκέφτομαι τη Σύρτη όπου γεννήθηκε ο Καντάφη και φυσικά όλος αυτός ο πληθυσμός που ουσιαστικά ήταν σαν καταραμένος ε, ήταν ε, κοντά στον Καντάφη αποκλείστηκε και έτσι αμέσως αναζήτησε ένα νέο πολιτικό εταίρο που να του παράσχει κάποιο χώρο στην πολιτική ζωή. Ε, αναρωτιέμαι λοιπόν αυτή η υποστήριξη που δώσαμε σε κάποιες κυβερνήσεις Αλμαλή στο Ιράκ ε, στην μεταβατική ε, κυβέρνηση της Λιβύης που ήταν ακόμη πιο εύθραυστη και που δεν κατάφερε να επιτύχει τους στόχους που είχε θέσει ε, τον αφοπλισμό των ε, μαχητών. Γι' αυτό έχουμε σήμερα την Κεντρική Τράπεζα που πληρώνει ένα σωρό μαχητές. Σπαταλώντα τα ελάχιστα εισοδήματα που υπάρχουν ακόμα, απομένουν ακόμα από τι πόλει πετρελαίων. Δεν μπορούμε λοιπόν να αποκομίσουμε κάποια ε, διδαγμάτα από τι θέσει που κρατήσαμε κατά τη μεταβατική φάση. Και θεωρώ εμεί ω Ευρωπαίοι δεν θα έπρεπε να εμπλακούμε λίγο περισσότερο με κάποια δομή γιατί ξέρετε η Λιβύη βγαίνει από 42 χρόνια δικτατορίας είναι μια εύθραυστη χώρα ε, διάφορες φυλές υπάρχουν αστάθεια μεταξύ των διαφόρων φατριών δεν μπορούμε μόνο να τους πληρώνουμε δεν θα έπρεπε να συμμετέχουμε και κάπως πιο ενεργά σε αυτή τη μεταβατική διαδικασία τώρα όσον αφορά τα εσωτερικά προβλήματα της τρομοκρατίας. Θεωρώ ότι ένα από τα αίτια είναι κάποια προβλήματα που δεν αντιμετωπίσαμε αρκετά. Σκέφτομαι στην Βόρεια Αφρική οι περισσότερες κοινότητες ε, ανήκουν ε, στη σχολή ε, Μαλική της είναι η πιο αρχαία σχολή, πιο ανοιχτό μυαλή όσον αφορά την ερμηνεία και με μεγαλύτερη ενοχή. Αντιθέτως κάποια κράτη του κόλπου τις τελευταίες δεκαετίες ε, ε, προχώρησαν σε μια ερμηνεία πιο συντηρητική όπως οι Βαχαμπίτες. Ε, δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχουν συνέπειες μεταξύ σαλαφιστών και Βαχαμπιστών αλλά ε, σε αυτή την προσπάθεια αντικατάστασης ε, των παλιών συνετικών σχολών με τους Μαχαμπίτες ε, ανοίγεται μια οδός για κάποιους πιο ευάλωτους πληθυσμούς για κοινωνικούς, οικονομικούς λόγους έτσι λοιπόν αυξάνεται ο κίνδυνος ριζοσπαστικοποίησης μήπως θα έπρεπε λοιπόν και εμείς να αλλάξουμε στάση ως προς αυτά τα προβλήματα απαιτώντας ώστε όλοι αυτοί που υποστηρίζουν ε, αυτές τις απόψεις ε, να συνάδουν ε, κάπως να συμμορφώνονται με τις δημοκρατικές αξίες που χαρακτηρίζουν τις χώρες μας. Για τη Λιβύα το είπατε πολύ σωστά. Το έχω πει συχνά στην Ολομέλεια αυτά. Αποτελεί περισσότερο πρόβλημα παρά λύση. Πρόκειται για ένα άτομο που δεν κρύβει τη φιλοδοξία του να γίνει ο νέος Καντάφη, ένα αυταρχικό, ένας αυταρχικός πρόεδρος ε, και δεν είναι και κανένας μεγάλος στρατάρχης. Ε, ε, το βιογραφικό του στο στρατικό τομέα δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο και επιπλέον σήμερα προσπαθεί να παρεμποδίσει τη διαδικασία συμφιλίωσης, επανένωσης τα καταφέρνει σε κάποιο βαθμό γιατί κάποιε χώρε του το επιτρέπουν. Ε, και αναφέρομαι τώρα στην Αίγυπτο που έχει κάποιες ε, φιλοδοξίες ε, και που θέλει και κάποιον οικονομικό έλεγχο των πετρελαϊκών πόρων αλλά αναφέρομαι και στη Γαλλία αυτό που διαβάζουμε στον τύπο η οποία στέλνει ειδικέ δυνάμεις εκεί στην Κυριναϊκή που ενδιαφέρει επίσης και την Αίγυπτο, ώστε να συνεργαστούν με τις δυνάμεις του αυτά για να ε, καταλάβουν περισσότερο εδάφη. Αυτές οι προσεγγίσεις λοιπόν επιτρέπονται σε εποχές όπου γίνεται αυτή η προσπάθεια του ΟΗΕ και που είναι εύθραυστη και μια κυβέρνηση που, ε, όπου δεν υπάρχει πραγματικός έλεγχος και εξουσία. Δηλαδή οι ευρωπαϊκές χώρες και οι σύμμαχες χώρες ε, δεν θα έπρεπε να δείχνουν κάποια συνοχή και δεν θα έπρεπε να απορρίπτουν την προσωπικότητα του Αφτάρ, ο οποίο είναι επικίνδυνος ε, και για το θέμα της τρομοκρατίας πρέπει να πω γιατί παρουσιάζεται ο σύμμαχος της Δύσης αλλά εγώ διαφωνώ κάπως με αυτή την άποψη. Και μια τελευταία ερώτηση. Έχουμε την Αλγερία, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο. Έχει τεράστια έκταση, πολύ μεγάλο πληθυσμό, αλλά είναι σημαντική και για άλλους λόγους. Η τιμή του πετρελαίου, έτσι όπως έχει σήμερα, ε, οδηγεί στο ότι η αλγερινή οικονομία δεν είναι βιώσιμη, οπότε υπάρχει κίνδυνος ε, να δημιουργηθούν ε, κάποιες συνθήκες δυσαρέσκειας, θυμού στον αλγερινό πληθυσμό, ένα λαό πολύ παλιό και που χαρακτηρίζεται από γεροντοκρατία θα έλεγα. Οπότε μήπως μέσα στα επόμενα χρόνια υπάρχει κίνδυνος για νέο εμφύλιο πόλεμο ή κίνδυνος ε, ε, πραξικοπήματος που θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει ακόμη περισσότερο την περιοχή και να βρεθεί την Ισία μεταξύ μιας Λιβύης και μιας Αλγερίας ε, και να πέσει το χάος. Τι μπορούμε να κάνουμε κατά την άποψή σας για να αποφύγουμε μια τέτοια ρήξη και να διευκολύνουμε τη μετάβαση. Ελπίζουμε σε πιο δημοκρατικά καθεστώτα σε χώρους όπως η Αλγερία. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα και εγώ να αναπτύξω λίγο τις προηγούμενες ερωτήσεις μου. Ε, υπάρχουν κάποιες αλλαγές που είναι σημαντικές από γεωπολιτικής άποψης και αφορούν τη, σκηνο... και τη Σουνητική κοινότητα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, γιατί ίσως δεν είναι τόσο σημαντικό το θρησκευτικό στοιχείο, όσο οι φιλοδοξίες που έχουν οι διάφοροι εμπλεκόμενοι. Αν δούμε την κατάσταση στο Ιράκ, και μία από τις πρώτες σας ε, παρατηρήσεις, κυρία Γκάου, ήταν η ανάγκη η κοινότητα να ενταχθεί στην πολιτική διαδικασία. αφού άλλωστε γνωρίζουμε την ε, επιρροή του Ιράν σήμερα και τι σχέσεις που έχει η κυβέρνηση του με τις άλλες χώρες αλλά και τις ειδικέ δυνάμεις της χώρας. Υπάρχουν πολλές εντάσεις ε. Υπάρχουν ε, σημεία έντασης και πεδία μάχης ακόμη. Ακόμα και όταν το Ιράν συμμετείχε στη συμμαχία για την καταπολέμηση του Ισλαμικού κράτους στη Συρία, είχαμε την ε, επιρροή της Σαουδικής Αραβίας και μέχρι πρόσφατα, μέχρι το πόλεμο δηλαδή, μέχρι την εποχή που έγινε ο πόλεμος στη Συρία, η Σουνητική κοινότητα κυριαρχούσε. Ήταν ε, νομίζω η μεγάλη πλειοψηφία οι Σουνίτες και υπήρχε η Χεσμολάχ από τη μία πλευρά, τα κράτη όπως το Ιράν. Ε, δηλαδή υπάρχουν αλλαγές, υπάρχει και η γεωπολιτική διάσταση. Ευχαριστώ. Ναι, θα ήθελα να σας ακούσω και τους δύο. Αλλά πρώτα απαντήστε κυρία Γκάουπ στον κύριο Καστάλντο που έκανε την τελευταία ερώτηση. Πολλά σχόλια θα προσπαθήσω να κάνω μια σύνοψη για να απαντήσω στα θέματα που αναφέρατε. Πρώτον, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αναδόμηση μετά από μια διένεξη και η σταθεροποίηση είναι μια δραστηριότητα που δεν γνωρίζουμε καλά και δεν έχει ερευνηθεί και ιδιαίτερα. Φυσικά είχαμε τη Γερμανία του 45 και όλα αυτά αλλά η ιδέα ότι εξωτερικοί παράγοντες μπορούν να συμβάλλουν σε μια σταθεροποίηση μετά από μια διένεξη είναι ιδέα που ε, γεννήθηκε τη δεκαετία του 80 περισσότερο. Και όπως είπατε κι εσείς, ε, η διεθνής κοινότητα γενική ε, δεν έχει χειριστεί καλά το Ιράκ, τη Λιβύη, αλλά και άλλες περιπτώσεις. Οι βασικοί λόγοι είναι μια πολιτική κόπωση μία ε, έλλειψη βούλησης ε, και απαρεμβόλη. Θυμηθείτε τον Οκτώβριο του 2011 όταν η Λιβύη αρνήθηκε οποιαδήποτε παρέμβαση από το εξωτερικό. Και εμείς χαρήκαμε βέβαια που οι Λιβύοι θέλησαν να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους. Σήμερα χρειάζεται μια προσέγγιση πρώτα απ' όλα επικοδομητική. Δηλαδή να έχουμε μονίμως κάποιους στόχους, κάποιους μακροπρόθεσμους στόχους και να υπάρχουν, συμμετέχουν και όλοι οι διεθνείς εταίροι, να υπάρχει μια καλή συνεργασία που δεν υπήρξε μέχρι στιγμής και να δούμε και ποιοι βλάπτουν. Τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει διαφορετικά το 2011 στη Λιβύη, δηλαδή ο ΙΕ θα μπορούσε να έχει στείλει μια αποστολή επιτόπου, μια μικρή αποστολή η οποία θα είχε αφοπλίσει τους ε, ενόπλους, αλλά δεν ήταν η κατάλληλη πολιτική στιγμή. Δεν υπήρχε πολιτική βούληση ούτε από πλευράς Λιβύης, ούτε από πλευράς διεθνούς κοινότητας. Η ε, ασφάλεια τέθηκε σε πρώτο επίπεδο και μετά η οικονομία. Οπότε εμείς χρειαζόμαστε περισσότερη έρευνα στον τομέα αυτό, ώστε όπως είπα προηγουμένως να μπορούμε να δώσουμε μια εντολή στους πολιτικούς, να λάβουν οι πολιτικοί μια εντολή από τον πληθυσμό ε, βάσει του επιχειρήματο ότι θα είναι πιο αποτελεσματικό το να κάνω κάτι τώρα παρά να περιμένω μια πενταετία. Ε, είναι κάτι που πρέπει να δούμε κι εμείς ε, στο απόψη έρευνα, Ναι, να συμμετέχουμε περισσότερο, αλλά με τρόπο που ονομάζεται local ownership και μακροχρόνια, δηλαδή μια δεκαετία τουλάχιστον, διότι δυστυχώς με το Twitter και το Facebook όλα κινούνται τόσο γρήγορα που ο Ευρωπαϊκό πληθυσμό, άμα του ζητήσει κανεί μια εντολή δεκαετή, ε, δεν πρόκειται να την δώσει εύκολα. Για το Χαφτάρ ε, και για την ασφάλεια στη Λιβύη. Πιστεύω ότι οι χώρες που βρίσκονται επί τόπου το κάνουν περισσότερο για θέματα ασφάλεια όσον αφορά τον ΤΑΕΣ. Αλλά πράγματι, το είπα και προηγουμένω, χρειάζεται μια πιο μακροχρόνια και μια πιο ολιστική προσέγγιση Στη Λιβύη δεν μιλάμε για μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας, αλλά ανοικοδόμηση, γιατί ό,τι μένει δεν είναι και πολύ. Και ο Χαφτάρο, όπω είπα προηγουμένω, που ισχυρίζεται ότι είναι στρατάρχης ενός στρατού, δεν είναι στρατός πραγματικά αυτός, μιλάμε για 5-7 άτομα. Ε, και συμφωνώ στα όσα είπατε για την προσωπικότητά του και το ρόλο του. Ε, τέλος, ε, Αλγερία. Έχουμε συζητήσει αρκετά πρόσφατα για την Αλγερία. Συμφωνούμε κάπου με τις δικές σας ανησυχίες. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι αυτό θα γίνει σύντομα ούτε εμφύλιος πόλεμος, ούτε κάτι βίαιο άλλο. Αλλά σίγουρα εισέρχεται σε μια φάση μετάβασης πολιτικής η Αλγερία αλλά μετάβασης και αλλαγής γενιάς. Έχουμε μια νέα πολιτική γενιά που αφήκνεται τώρα πώς οι ηγέτες θα διαχειριστούν όλη αυτή την κατάσταση. Εγώ προσωπικά από την εμπειρία μου με τους Αλγερινούς πιστεύω ότι το σύστημα τους δεν είναι ιδεολογικό. Είναι αρκετά ε, επικεντρωμένο στην αποτελεσματικότητα. Οπότε δεν είμαι τόσο όσο εσείς. Ε, αλλά είναι σαφές ότι πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί οι διαβλοί επικοινωνία. Η Αλγερία είναι μια χώρα με μεγάλη υπερηφάνεια και εμεί ω Ευρωπαίοι δεν έχουμε δυνατότητα να επηρεάσουμε οτιδήποτε στην Αλγερία. Πρέπει να συνεχίσουμε τι συναλλαγές, την οικονομική συνεργασία και να παίξουμε ένα ρόλο σημαντικό όπω και στη Λιβύη και στην Τινησία, αλλά η οικονομική κατάσταση δεν έχει φτάσει ακόμη στο σημείο όπου υπάρχει κίνδυνο για κατάρρευση με στο επόμενο έτος. Είναι λίγο ανησυχητικά δηλαδή τα πράγματα, αλλά όχι ε, υπερβολικά. Να κλείσω λιγάκι τη συζήτηση αυτή σε σχέση με την αντιπαράθεση των ΣΥΙΤΟΝ με τους Σουνίτες. Όπως είπατε δεν είναι θέμα μονάχα σεκταρισμού, είναι και τα εθνικά συμφέροντα των δύο χωρών που είναι οι κύριοι παίκτες στη Μεσανατολή της Σαουδικής Αραβίας και το Ιράν. Αν δούμε τις Ιρανικές δράσεις τα τελευταία δέκα χρόνια, βλέπετε ότι προσπαθούν να προστατεύσουν τα συμφέροντα των Σιητικών κοινοτήτων σε όλες τις περιοχές της Μέσης Ανατολής. Αν δείτε το δυτικό τμήμα του Αφγανιστάν, παραγωγός χάρη, το Αζερβαϊτζάν, τη Συρία, τη Λιβύη, το Μπαχρέιν, την Ιεμένη, σε όλες τις περιπτώσεις που έχει δράσει το Ιράν, είναι ουσιαστικά η προστασία των συμφέροντων της Σιητικής κοινότητας. Το καλό νέο είναι τώρα ότι μετά από την άρση των κυρώσεων εναντίον του Ιράν, η εξωτερική πολιτική του Ιράν άρχισε να γίνεται πιο θετική, γιατί δεν χρησιμοποιούν πια την ε, ήπια δύναμή τους στον Κάφκασο, στον Νότιο Κάφκασο όπως στο παρελθόν. Γιατί στο παρελθόν όταν οι Ιρανοί θεωρούσαν τους περιστοιχίζουν εχθρικά κράτη, εθνικές δυνάμεις προσπαθούσαν να ασκήσουν πραγματική εξουσία εξ ονόματος των σιητικών κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο. Βλέπουμε τώρα να μειώνεται η παρουσία τους και στο Γεωργία και στο Αζερβαϊτζάν γιατί δεν νιώθουν την ίδια εχθρότητα από τις χώρες αυτές. Δεν μπορούμε να πούμε ακριβώ το ίδιο βέβαια για τη Μέση Ανατολή γιατί η εξεράγη κατάσταση στην Ιεμένη, υπήρξαν τα προβλήματα στο Μπαχρέιν και φυσικά έχουμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Συρία και στο Λίβανο που είναι πάρα πολύ ενεργή στο δυτικό τμήμα του Αφγανιστάν. Εκεί υπάρχει σημαντική ιρανική επιρροή και ελέγχει μεν την περιοχή αυτή η κυβέρνηση του Αφγανιστάν, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη ήπια δύναμη εκεί το Ιράν. Πάρα πολλά πράγματα θα εξαρτηθούν από την απόλυξη αυτής της διαμάχης Σιητών και Σουνιτών, αν το Ιράν και η Σαουδική Αραβία θα συμφωνήσουν για τις σφαίρες επιρροής και ήπιας εξουσίας κάθε μίας από τις ε, δύο ε, χώρες και δεν θα μπουν ο ένας στα χωράφια του άλλου. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε εδώ αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους δύο διακεκριμένους ομιλητές για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστώ και όλους εσάς που συμμετείχατε και παρακαλώ να έρθετε και το απόγευμα που έχουμε αυτή την κοινή ακρόαση, πολύ ενδιαφέρουσα μεταξύ, μεταξύ ΣΕΝΤΕ και ΛΥΜΠΕ. Ε, με θέμα διασφάλιση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι με μας, την Επιτροπή μας και την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνη και Εσωτερικών Υποθέσεων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι μια πρόκληση για την εξωτερική και εσωτερική ασφάλεια. Ελπίζω ότι θα έρθετε. Ευχαριστώ πολύ.